Uh, So good morning, everybody. I think um, I'm just going to make my opening announcements because we're waiting for our rapporteur to um, to arrive to start the exchange of views on our first item, which is an opinion. Να κάνουμε την ανταλλαγή απόψεων και το πρώτο σημείο, πρώτα απ' όλα, γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερο, επανεκβιομηχάνηση της Ευρώπης είναι το πρώτο σημείο. Σας το λέω. Επειδή δεν είμαστε πολύ σημαντικά θα αίθουσα, μεγάλη αίθουσα όμως στη διάθεσή μα, γιατί το απόγευμα υπάρχει μια πολύ σημαντική ακρόαση για την ιστορική αγορά των υπηρεσιών. Η κυρία Βίλιτσα. και η έκθεσή της για το πώς επηρεάζονται τελικά οι υπηρεσίες από το νέο πακέτο για την ανάπτυξη. Είναι το αντικείμενο που θα το απόγευμα και σας ενθαρρύνω να διαβάσετε τα σχετικά έγγραφα. Επίση να καλημερίσω όσου μας παρακολουθούν μέσω web streaming. Επίσης, σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει και το μηνιαίο newsletter που ε, μόλις δημοσιεύθηκε. Αν δεν το έχετε λάβει στο mailbox σας, υπάρχει και ένα email στην πέσω σελίδα και μπορείτε να μας στείλετε το email σας. Ήδη έχουμε 2.000 συνδρομητές μέσω email για να σου στείλουμε. Και Υπάρχει μια ομάδα επικοινωνία στο Κοινοβούλιο που ε, μας στέλνει ιδέες και εμείς έχουμε κάποιες ιδέες για να βελτιώσουμε όσο γίνεται καλύτερο ε, τον τρόπο που επικοινωνούμε τη δουλειά μας. Ως ουσιαστικά επαγγελματικό δίκτυο για κάποιες ε, δραστηριότητες business to business. Πρώτα απ' όλα, θέλω να πω ότι θητούμε επισήμως την ημέρα διάταξη από τους παρόντες Βλέπω ακριβώς Πρότσερ και κυρία Μίλλερ πολύ πολύ μακριά σε αυτή την αίθουσα από μένα. Έτσι έχουμε λιγάκι καθίσει δυσπραμένα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη σε διάταξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν μου επιτρέπετε να σας παρουσιάσω τις εντατικές εργασίες που έχουμε αυτό το δίμερο. Αύριο θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις για μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση για τις κλινικές δοκιμές. Και πολλές αποφάσεις πρέπει να πάρουμε επί διαδικασιών για πολύ σημαντικές νομοθετικές προτάσεις που αυτή τη στιγμή διεκπαιρώνει το σύστημα σε ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες κτλ. Όπως επίσης έχουμε τη γραμμοδότηση για την απόσπαση εργαζομένων. Στις 10 και 4 ο κύριος Μπαρνιέ θα είναι μαζί μας να μας πει λίγα λόγια για τα σχέδιά του για το, τη τελευταία πλήρη χρονιά που έχουμε ε, μπροστά μας ε, όλοι εδώ. Και από τα κύρια Γκέπα, ο κύριος Χάνς Πίτερ Μάγερ θα μας ενημερώσουν για το έργο του Κοινοβουλίου για τη μελέτη για το Ευρωπαϊκό Νόμο Πολύσεων. Πολύ σημαντικό θέμα και θα ξεκινήσουμε κατά απόγευμα μια συζήτηση για πολύ σημαντικέ πρωτοβουλίε όπω η ηλεκτρονική ταυτοποίηση και υπηρεσίε εμπιστοσύνη για τι ηλεκτρονικέ συναλλαγέ στην ιστορική αγορά. Πολύ βεβαρημένη μερική διαταξή λοιπόν. Αυτά από πλευρά μου. Εκτό αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Οπότε να καλημερίσω και να καλωσορίσω την κυρία Γκεφάρτ, τη συγγήτριά μας και να την καλέσουμε να παρουσιάσει τη γνωμοδότησή για την εκμηχάνηση της ε, ε, Ευρώπης. Και αυτό ε, έρχεται ως απάντηση στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη θέματα αγωνιστικότητας και βιωσιμότητας, κάτι πολύ σημαντικό για μας. Θα δώσω το λόγο μέσω στην εισηγήτρια. Ο κύριος Φαπ θα μιλήσει εξ ονόματος της κυρίας Κρέμη. Ο κύριος σε ονομάτως του κύριου, του κύριου Χάζη Μαρκάκη. Άλλο τους θα πάρουν το λόγο, έτσι δεν είναι. Η κυρία Ρούλερ είναι παρούσα. Εγώ θα μιλήσω σε ονομάτως της ομάδας μου και οποιοδήποτε άλλος επιθυμεί να συμμετάσχει στη συζήτηση με χαρά. Για να μην καθυστερώ πρατερό, κυρία Κέχαρτ, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και χαίρομαι για την ευκαιρία αυτή τη συζήτηση, έστω και δεν είναι παρόντε οι περισσότεροι σκιώδης ηγητές. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολύ αξιόλογη. Γιατί έχουμε εμπειρία και λόγω της ε, οικονομικής κρίσης. Έχουμε διαγνώσει ότι δεν ε, λειτουργούν πολλά κομμάτια της εσωτερικής μας αγοράς όπως θα έπρεπε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι, αν θέλουμε μια καλύτερη παρουσία στην πολιτική αλλά και την οικονομία, μάλλον αν είχαμε μια καλύτερη παρουσία στην πολιτική και την οικονομία, ε, ίσως να αντιμετωπίζαμε πιο ευχερό στην κρίση, να ήταν λιγότερο βαριές οι της από ότι τώρα. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να επισημάνω ότι τα ζητήματα πολιτικής που έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες ήταν αυτά τα οποία πλήξαν περισσότερο από την κρίση. Γι' αυτό και θεωρώ ευπρόσδεκτη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και την εστίαση στον συστήσεων μας αυτή. Χρειάζεται μια βιομηχανική πολιτική αποφασιστική με προγραμματισμό που να καλύπτει πολλούς τομείς πολιτικής, γιατί δεν είναι μόνο οικονομική πολιτική, βιομηχανική, δεν είναι μόνο δημοσιονομική, δεν είναι μόνο αυτά, είναι ακόμη και κοινωνική αλλά και περιβαλλοντική πολιτική, η πολιτική για τη βιομηχανία. Και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση, μια γενική προσέγγιση. Δεν θα επαναλάβω τις ε, παρατηρήσεις μου, τα έξι σημεία στα οποία έχω επικεντρωθεί. Ασφαλώ μπορούν να τα αναγνώσουν οι συνάδελφοι και οι πολίτε εφόσον ενδιαφέρονται, μπορούν να τα αναζητήσουν στο ίντερνετ. Θα ήθελα μια και δεν έχουμε πολύ χρόνο να επικεντρωθώ σε αυτά που ε, δεν είχα χώρο στην έκθεσή μου, στη γνωμοδότησή μου να περιλάβω, αλλά που πιστεύω ότι μπορούμε χάρη στις τροπολογίες να συμπληρώσουμε. Ξεκινώ λέγοντας ότι Η γενική βάση της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον άρχισα να με κατέπληξε, διότι εγώ ε, σε κάποια σημεία έβλεπα να μιλάει για προγραμματισμένη οικονομία. Διότι αναφέρονταν συγκεκριμένοι τομείς βιομηχανικής δράσης για τους οποίους θα έπρεπε να προσφερθεί ειδικά η στήριξη. Και σε αυτό θα πω ότι δεν είμαι βεβαία πως πρόκειται για το σωστό δρόμο. διότι η βιομηχανική, επιτροπή, η ε, βιομηχανική ε, πολιτική, ιδιαίτερα σε χώρες όπως μας που βρίσκονται σε ανταγωνισμό ευθύ με την Ινδία και την Κίνα, δεν μπορεί να έχει ανταγωνιστικότητα στους παραδοσιακούς τομείς της βιομηχανίας. Χρειαζόμαστε καινοτομία, χρειαζόμαστε νέες λύσεις, τεχνολογία εχμής πάνω απ' όλα. Και παρόλα αυτά σήμερα ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιες... Ε, καινοτομίες θα έχουμε μπροστά μας αύριο, μεθαύριο, στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι πολύ ε, ευχαίρες να διατυπώσει κανείς συγκεκριμένε προτάσεις. Εγώ αυτό που προτείνω είναι ιδιαίτερα να δώσουμε έμφαση στην καινοτομία, την έρευνα, την ε, απόκτηση δεξιοτήτων μέσα από το, από, από το Πανεπιστήμιο, ώστε να στελεχώσουμε μια ε, βιομηχανική δράση, μια έρευνα και τεχνολογία που μακάρι να φέρει και βραβεία Νόμπελ στο μέλλον στην Ευρώπη. Αλλά επαναλαμβάνω δεν είναι δυνατόν να κάνουμε πρόβλεψη και προγραμματισμένη οικονομία σε τομείς για τους οποίους δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον. Ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό σε σχέση με αυτά που έκανε στην ε, ομιλία του προς το ε, έθνος όπως ονομάζεται ο Μπαράκ Ομπάμα που άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και ίσως θα μπορούσε να δώσει κάποιες ιδέες και για τους Ευρωπαίους. Στην ε, εν λόγω ομιλία λοιπόν ο Μπαράκ Ομπάμα υπεγράμμισε ιδιαίτερως δύο σημεία δύο σημεία που εγώ θεωρώ πολύ σημαντικά για τη βιομηχανική μας πολιτική. Ιδιαίτερα λοιπόν τόνισε τον ελάχιστο μισθό διανόμο ότι θέλει να τον ορίσει στα 9 δολάρια αυτό αποτελεί ένα σαφέ μήνυμα ότι μπορούν ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε με το μέσο αυτό, με το μέτρο αυτό να βοηθήσουν στην ανάπτυξη εσωτερική ζήτηση και ω εκ τούτου να βοηθήσουν στην αναζωογόνηση τη οικονομία. Και δεύτερον, σαφέ μήνυμα για ε, επαναβιομηχανοποίηση ε, και μια συμφωνία σχετική για σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένων Πολιτειών σε μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών. Αν ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία, μπορούμε πιστεύω να περιμένουμε ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς, γιατί βέβαια τις διαπραγματεύσεις ε, θα τις ε, αναπτύξουν ε, οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει λοιπόν εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε προσδιορίσει τις κατευθύνσεις που επιδιώκουμε, που θέλουμε να δώσουμε, τι περιμένουμε από αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και αυτό είναι ένα από τα σημεία που ήθελα να περιλάβω στην έκθεσή μου. Αλλά δεν μπορούσα να περιλάβω λόγω έλλειψη χώρου. Άλλωστε δεν είχα προλάβει κιόλα να ακούσω την ομιλία του Μπαράκ ε, Ομπάμα την εποχή που τις ημέρες που έδινα το κείμενό μου στη μετάφραση ακόμη δεν είχε εκφωνηθεί αυτή η ομιλία. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει ίσως να είναι και το πιο δύσκολο είναι ότι χρειαζόμαστε μια εναρμόνιση του φόρου των επιχειρήσεων. Δεν είναι δυνατόν στην Ευρώπη να εξακολουθούμε να επιτρέπουμε αυτόν τον ε, κακό ανταγωνισμό, τον μη υγιή ανταγωνισμό μεταξύ κρατών μελών, που προσπαθούν να προσελκύσουν το καθένα στην επικράτεια του επιχειρήσεις. Διότι αυτού του τύπου ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών οδηγεί τελικά στην δημιουργία θέσεων εργασίας σε ένα κράτος μέλος εις βάρον άλλων θέσεων εργασίας σε άλλο κράτος μέλος. Δεν μπορεί να είναι αυτή η πολιτική μας για την οικονομία, για τη βιομηχανική δράση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε τις βέλτιστες προϋποθέσεις πλαισίου για τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε εν τέλει να ε, εξασφαλιστεί ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και όχι ανταγωνισμός αθέμητος μεταξύ των συστημάτων των κρατών μελών. Ξέρω πόσο ακαρθώδες είναι το ζήτημα αυτό, αλλά ωστόσο θεωρώ ότι οφείλω να το φέρω στη συζήτηση. Επίσης βλέπουμε ότι αυτή η στρέβλωση του ανταγωνισμού ως προς ε, τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης που προξενείται από αυτή τη διαφορά στη φορολόγηση των επιχειρήσεων οδηγεί παραδείγματι την Κύπρο και την Ιρλανδία στο να αναπτύσσουν μία σειρά από επιχειρήσεις που ε, ε, ε, αναπτύσσουν την έδρα τους εκεί, δημιουργούνται εκεί, χωρίς όμως να έχουν βιομηχανική δραστηριότητα. Είναι μόνο επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Πού πήγε το τσάι μου, πού πήγε ο καφές μου. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα ήταν κακό ίσως να φροντίσουμε να δώσουμε καλύτερες λύσεις συνεργατικές και νομίζω ότι αυτό οφείλουμε να το συζητήσουμε. Μα εγώ ήθελα τσάι, δεν ήθελα καφέ. Μου πήρανε το φλιτζάνι μου, μου φέρανε καφέ χωρίς να τον έχω ζητήσει. Θα προτιμούσα τσάι. Εν πάση περιπτώσει, έστω. Και ε, πάω εδώ Ασφαλώς υπάρχουν και άλλε παρατηρήσεις που θα ξέρω τον κόπο να ακουστούν, αλλά α ξεκινήσει η συζήτηση, α μην μονολογώ εγώ. Και εν τέλει, μια και θα με ρωτήσει τόσο άλλο ο πρόεδρος στο τέλος, για το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα λοιπόν έχουμε τη συζήτηση προθεσμής για την κατάθεση των τροπολογιών στις 26 Φεβρουαρίου, στις 12 το μεσημέρι και προτείνουμε τη συζήτηση για τις τροπολογίες να τη δεξαγάγουμε στις 20 Μαρτίου, να γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή μας στις 24 Απριλίου και στην Επιτροπή Βιομηχανίας τον Μάιο του 2013 πάντα. Ελπίζω ότι μπορούμε έτσι να ε, εργαστούμε χωρίς υπερβολική χρονική πίεση και ε, περιμένω την πολύ καλή συνεργασία με τις και τους χειώδεις συγκητρίες και συγκητές και την ε, ολοκλήρωση της δουλειάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύ καλή σας παρουσίαση και έχετε προσθέσει και νέα τροφή για σκέψη με την παρουσίασή σας. Εγώ για πρώτη φορά θα συμμετάσχω σε έναν, ε, μια υπερατλαντική, αν θέλετε, ομάδα ε, συζήτηση και διαπραγματεύσεων ε, ευρύτερα για την βιομηχανική πολιτική, για πρότυπα, χωρίς ε, εμπόδια, που είναι κάτι που μας ζήτησε η Αμερικανική Αντιπροσωπεία να συζητήσουμε και ελπίζω να καταφέρουμε κατά τη διάρκεια των, ε, της συναδρίας των συντονιστών να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη διαδικασία καθώς η Επιτροπή μας έχει μεγάλο ε, ρόλο να διδραματίσει λόγω της εμπειρίας της σε τέτοια ζητήματα. Άντες Φάρμπ, έχετε το λόγο. Εκ μέρους του ΕΛΚ. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. καθιστώ εγώ εδώ την κυρία Κόμε, τη συνάδελφο που είναι ισχυώδης για τη γνωμοδότηση αυτή και κάποιες ε, πολύ σημαντικές υποχρεώσεις στην Ιταλία και δεν μπόρεσε να έρθει. Με παρακάλεσε όμως να την εκπροσωπήσω και ξεκινώ λέγοντας ότι συμφωνεί σε πολλά σημεία της γνωμοδότησης, το κείμενο που έχει. Στο σημείο 4 η, η συντάκτρια προτείνει έναν ε, ελάχιστο μισθό στην ε, βιομηχανική πολιτική. Και σε αυτό θα παρατηρήσω ότι Ακόμη και αν όλα τα μέλη τη Επιτροπή μα ή η πλειονότητα των μελών τη Επιτροπή μα συμφωνήσουν στην πρόταση αυτή, είμαι βεβαίω ότι η Βιομηχανική Επιτροπή δεν θα συμφωνήσει καθόλου στο να μπαίνουμε στα δικά τη χωράφια. Εδώ τώρα θα ήθελα να προσθέσω μία παράγραφο που πιστεύω θα μπορούσε να οδηγήσει στη βελτίωση των, ε, της αγοράς αγαθών ε, προϊόντων δηλαδή στην Ευρώπη. Γιατί ξέρετε υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία παράγονται και είναι πολύ καλής ποιότητας, παράγονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να καταναλώνονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω θα πρέπει να προσθέσουμε μια σχετική παραγραφή. Και βεβαίω η αγορά για τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελεί ένα σοβαρό σημείο και πρόβλημα σε σχέση με την πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν έχει καλύψει. Ο τομέα τη Άμυνα και των εξοπλισμών που πολλέ φορέ μα έχει απασχολήσει από την αρχή τη θετίας μα. και εν τέλει θα πρέπει να δούμε εάν θα περιλάβουμε κάτι για την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης ως προς την ασφάλεια και ποιότητα των βιομηχανικών προϊόντων. Η ομάδα μας δέχεται μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική σαν Πιστεύουμε ότι έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα στη μηχανική παραγωγή στην Ευρώπη και πρέπει να τα αναπτύξουμε. Ο τομέα των υπηρεσιών και ε, από μόνο του δεν μπορεί να δώσει λύσει στα προβλήματα του. Αντίον θα επιδεινώσει την κρίση στην Ευρώπη και ο ανταγωνισμό δεν επαρκεί. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε έμφαση στην βιομηχανική μα πολιτική και να λάβουμε τι απαραίτητε αποφάσει. Η κύρια πιο σημαντική απόφαση είναι για τις βιομηχανίες πλαισίου της ε, λειτουργίας της βιομηχανίας στην Ευρώπη. Να δώσουμε λύσεις που θα τις βελτιώσουν, χωρίς πάντα να είναι πολύ κακές που πρέπει να βοηθήσουμε να βελτιωθούν, διεξόδους και ως προς την δραστηριότητα, θέματα παραδείγματι που έχουν να κάνουν με την περιβάλλον που όμως ωστόσο θα πρέπει η Επιτροπή Περιβάλλοντος να εξετάσει, αλλά στα οποία θα πρέπει εμείς να δώσουμε την έφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί χρειάζονται ειδική μεταχείριση. Και εν τέλει, για να καταλήξω, ε, συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με τα όσα καταγράφονται στη γνωμοδότηση. Η κυρία Κόμη, και οδησηγήτρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα κάνει βεβαίως κάποιες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Χατζημαρκάκης έχει το λόγο. Um, äh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ θα συμφωνήσω Συμφωνώ και εγώ με την ε, κυρία Γκέπχαρτ σε πολλά σημεία. Το σημείο 4 που έθιξε και ο κύριος Σφαπ μας δίνει έναν χαρακτηριστικό τόνο θα έλεγα για τη γνωμοδότηση, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι είναι θα το λύσουμε τις τροπολογίες. Θα ήθελα προκειμένου να υπογραμμίσω ότι η βιομηχανική παραγωγή και το είπατε και εσείς ε, και ο κύριος Σφαπ αποδυναμώνεται διαρκώς στην Ευρώπη και όχι μόνο σε κάποια κράτη που είχαν δασική βιομηχανική παραγωγή, αλλά ανά την Ευρώπη. Εν γέννη παρατηρείται ότι η παραγωγή, ακόμη και η μικρής κλίμακα βιομηχανική παραγωγή, ε, επικεντρώνεται σε ορισμένα αστικά κέντρα ή περιορισμένα αστικά κέντρα και εν γέννη η περιφέρεια και η ύπεθρος υποφέρει σημαντικά και βρίσκεται σε δυσμενή θέση και λόγω της Εσωτερική αγορά, διότι φαίνεται ότι η εσωτερική αγορά έχει ενισχύσει του ισχυρού, αλλά έχει αποδυναμώσει του πιο αδύναμου αυτή την ιστορία. Και γι' αυτό πρέπει να αναλογιστούμε πολύ σοβαρά τη βιομηχανική μα πολιτική. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κράτη τη περιφέρειας όπω η Πορτογαλία, όπω η Ελλάδα αλλά και η Ισπανία έχουν, ε, παρουσιάσουν μια απόλυτη κατάρρευση της βιομηχανικής του διαδραστηριότητας και γι' αυτό θα πρέπει ίσως να αναζητήσουμε κάποια μέτρα που θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις. Εδώ βεβαίως πρέπει να συζητήσουμε τα συστήματα των, ε, της εκπαίδευσης στα κράτη που αποτελούν και ένα πολύ, εξαγωγη, ε, πολύ εξαγώγημο προϊόν μας ε, και ενώ εκπαίδευση όχι μόνο στο πανεπιστήμιο αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση που, ξεκινά, που συνεχίζει την πανεπιστημιακή μόρφωση, επαγγελματική κατάρταση, εκμάθηση για τους νέους, μέσα σε μια μικρή επιχείρηση. Στο πεδίο αυτό λοιπόν χρειάζεται ακόμη περισσότερη βελτίωση, γιατί εδώ μπορούμε να ε, πούμε ότι από αυτήν θα εξαρτηθεί και η ποιότητα του προϊόντος, η ποιότητα των αγαθών που παράγουμε και εξάγουμε. Ίσως και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο έχει τόσο καλές επιδόσεις η γερμανική, η αυτή τη στιγμή. Το δε σύστημα αυτό, το διαδικό όπως ονομάζεται, δηλαδή μόρφωση στο σχολείο και εκμάθηση ε, στην πράξη με την ε, πρακτική εκπαίδευση στη συνέχεια προσπαθεί και η Ισπανία τώρα να το εισαγάγει. Έτσι λοιπόν, καταρχάς πρέπει να γνωρίσουμε ότι δεν υπάρχει υποστήριξη σε ισότιμους όρους ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το κάθε κράτος επιλέγει τις δικές του λύσεις ε, οι οποίες εν τέλει δεν φέρουν συγκρίσιμα αποτελέσματα οι πολιτικές, οι ευρωπαϊκές πάλι δεν δίνουν αυτή την λύση που θα θέλαμε, την ε, εκτεταμένη υποστήριξη δηλαδή της βιομηχανίας και λύσεις μέσω είτε εθνικών είτε ευρωπαϊκών ε, τραπεζών βιομηχανικής ανάπτυξης. Και εδώ ιδιαίτερα θα πρέπει να δώσουμε Ε, έμφαση σε αυτές τις τράπεζες της ε, βιομηχανικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα για τα κράτη όπου δεν υπάρχουν και ίσως μπορούμε ε, όπου υπάρχουν αυτές τις τράπεζες όπως η ΚΑΕΦΕ η Γερμανική, η Τράπεζα για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη, να δραστηριοποιηθεί και σε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν αντίστοιχες αντίστοιχου οργανισμού υποστήριξη βιομηχανική δραστηριότητα. Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει επίση θα χρειαστούν ιδιαίτερη υποστήριξη, πάντοτε το επενθυμίζουμε. Ένα πρόβλημα σημαντικό εδώ είναι οι καθυστερήσει στι πληρωμέ, οι υπερημερίε. Ένα ζήτημα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε και να δώσουμε αποτελεσματικέ λύσεις στην Ευρώπη. Thank you Κυρία Ρούλα, Ευχαριστώ πολύ και πολύ στόμα γιατί καλύπτηθηκαν όλα. Ένα σημείο θα υπογραμμίσω μόνο. Συμφωνώ με την κυρία Γκέπχαρτ ότι δεν είναι δυνατόν η ε, κεντρική ε, ένα κεντρικό φορολογικό σύστημα να βοηθήσει την ανάπτυξη τη βιομηχανική δραστηριότητα. Αυτό δεν το καταφέρουν τα κράτη-μέλη, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνει. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει έμφαση στην έρευνα, στην τεχνολογία, την επιστήμη. Τώρα αυτό πώ ε, συνάδει με τι περικοπέ του προπολογισμού, ιδιαίτερα στο πολιτεύσιμο οικονομικό πλαίσιο, θα ήθελα να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν η κυρία Γκέπχαρτ έχει να πει δύο λόγια για αυτό, αλλά δεν είναι δυνατόν να το αγνοήσουμε το φαινόμενο αυτό. Πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε μια σχετική παρατήρηση μέσα στη γνωμοδότηση και κατά τα άλλα θα συμφωνήσω με τον κύριο Χατζημαρκάκη για τη διαδική μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση. Αλλά πρέπει να επισημάνω εδώ ότι αυτό το σύστημα δεν έχει φέρει τα απαιτούμενα αποτελέσματα ή τα αναμενόμενα αποτελέσματα ω προ την αναγνώριση των ισοτιμιών των πτυχίων. Και σε αυτό θα πρέπει να κάνει, ή των επαγγελματικών δεξιοτήτων καλύτερα, και σε αυτό θα πρέπει να κάνει μια προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Να πω και εγώ δύο λόγια, μετά να δώσω το λόγο στον συνάδελφο και σε οποιονδήποτε άλλο θέλω να πάρει το λόγο. Ο κ. Καπελέρο Σάνσα είναι δεκμένο τη Επιτροπή. Ε, τον καλωσορίζουμε. Συγγνώμη που δεν το έκανα προηγουμένω. Θα ακούσουμε και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον στο έγγραφο της Επιτροπής ε, για μια ισχυρότερη ε, βάση για την ευρωπαϊκή οικονομική ανάπτυξη είναι ότι πρώτα απ' όλα θα ήταν χρήσιμο και θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι αυτή η πρόταση έχει εξαιρετικά ισχυρέ συστάσει για την ενιαία αγορά, την εσωτερική αγορά. Και εδώ παραθέτω ότι είναι πολύ σημαντικό να διασκεδαστούν αβεβαιότητες στις νέες αγορές για ένα σταθερό και προβλέψιμο μακροπρόθεσμο πλαίσιο συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας. Αυτό είναι το πρώτο ε, στοιχείο που θα ήθελα να θέσω εδώ, σε αφορά την, τις επιχειρήσεις, είτε είναι βιομηχανία, είτε επεξεργασία. Μιλάμε για μακροπρόθεσμες επενδύσεις και έτσι θα χρειαστεί μια περίοδος εγκατάστασης, αγοράς εξοπλισμού, αλλά όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές αποφάσεις για τις επιχειρήσεις. για τέτοια ζητήματα μπορούν ε, να πάρουν πολύ καιρό να αποφασιστούν γιατί περνάνε από κοινοβούλια, περνάνε από επιτροπές και κάποιες φορές όταν εξετάζουμε αυτές τις ε, πολιτικές τη ε, ενιαία αγορά, δεν εξετάζουμε αυτές τις μεμονωμένες στοιχείες. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που θα ήθελα να τονίσω. Ευρύτερα όμω, θεωρώ ότι όλη η ισορροπία μεταξύ οικονομιών είναι σημαντική. Αναφέρθηκε ότι κάποιες χώρες που έχουν ισχυρό βιομηχανικό πυρήνα τα πάνε καλύτερα εν μέσω κρίσης από τι άλλες. Αυτό ισχύει γενικά, αλλά στη χώρα μου παρά το γεγονό ότι ακόμα παλεύουμε ε, να κατακτήσουμε μια καλή ε, οικονομική ανάπτυξη, έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μεγάλο αριθμό θέσεων εργασία στον ιδιωτικό τομέα, ε, το οποίο τίνει να συμβαίνει και, στον, και στις επιχειρήσεις υπηρεσιών και έτσι δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν κόσμο πιο γρήγορα. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασία, η ικανότητα πρόσληψης ε, νέων εργαζομένων είναι εξαιρετικά σημαντική. Όπως αναφέρθηκε από τον κύριο Φάρεψε προηγουμένω, από ε, αφορά την Επιτροπή Απασχόληση περισσότερο και όχι εμάς. Εγώ είμαι επιφυλακτικός ό,τι αφορά την εναρμόνιση στη φορολογία που αναφέρεται σε αυτή την πρόταση, γιατί δεν ξέρω ότι είναι δική μας αρμοδιότητα και δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε επί ζητημάτων ε, εναρμόνισης ε, τέτοιων φόρων, ούτε θα συμφωνήσουμε σε ό,τι αφορά τη δομή των ε, φόρων που συνδέονται με την απασχόληση. Γιατί οι χώρες που έχουν υψηλά ποσοστά φορολόγηση των εργοδοτών ή εργοδοτικών εισφορών σίγουρα αποθαρρύνουν τους επιχειρηματίες από και πάλι τονίζω τη σημασία της, ε, ε, των μακροχρόνιων θέσεων εργασία ε, στο πλαίσιο της βιομηχανικής πολιτικής, γιατί το χαρακτηριστικό μιας επιτυχούς βιομηχανικής πολιτικής είναι η δημιουργία τέτοιων θέσεων εργασίας. Και ε, στις κατασκευαστικές ή παραγωγικές βιομηχανίες λέμε ότι έχει μειωθεί η απασχόληση σχετικά, όμως η παραγωγή, η απόδοση έχει αυξηθεί. Γιατί υπάρχει καινοτομία, υπάρχει εξέλιξη, μειώνεται ο χρόνος ε, τοποθέτησης του προϊόντος στην αγορά. Και συνολικά στην απασχόληση τι συμβαίνει στην βιομηχανία. Πολλές από αυτές τις βιομηχανίες γίνονται και ε, επιχειρήσεις υπηρεσιών. Γιατί έτσι δημιουργεί... αυτό είναι τμήμα της δημιουργίας της αξίας του προϊόντος. Θα ήθελα να, ε, θα να αναφερθώ στη Ροζ Ροζ για παράδειγμα που έχουμε στατιστικά στοιχεία. Ε, εδώ και χρόνια λοιπόν παράγουν ε, ιδιαίτερα ακριβά και περίπλοκα προϊόντα. Αυτή τη στιγμή το 40% των δραστηριοτήτων τις χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες. Γιατί κατασκευάζει με ε, μηχανές, αλλά μετά τις διατηρεί, τις συντηρεί, τις ε, ε μεταβάλλει σε μηχανές ε, αεροπλάνων και το καθεξής. Και έτσι υπάρχει ένα σοβαρό κίνητρο για τον κατασκευαστή, τον παραγωγό του προϊόντος, να το καταστήσει αρκετά αξιόπιστο και λειτουργικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα είναι ακόμα πιο οικονοποιημένοι οι πελάτες Το ίδιο ε, ισχύει και σε άλλους τομεί, ε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει αυτή η σωστή ισορροπία. Και μετά στην απασχόληση δεν υπάρχουν αλλαγέ στη δομή της σε αυτές τις επιχειρήσεις. Κλείνοντας, μιλάμε βεβαίω για την οικονομία που αφορά τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. και ακόμα και ο ορισμός κάποιες φορές δημιουργεί προβλήματα. Χθες, για παράδειγμα, ήταν εδώ το ε, Φόρουμ Επιχειρηματιών της ε, Μάλτας ε, και όσοι είχαμε πάει στην ε, Κύπρο και εκεί είχαμε κάνει εκτενείς συζητήσει για τη δομή της οικονομίας. Και οι δύο αυτές οι οικονομίες βασίζονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όπως και οι Μαλτέζοι μου υπέδειξαν, μια επιχείρηση που απασχολεί 150 ε, εργαζομένους ε, που χαρακτηρίζεται ως μικρομεσαία επιχείρηση στη Μάλτα είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε τις ε, διάφορες δομές που μπορεί να λάβει μια οικονομία γιατί φαίνεται ότι οι νέες τεχνολογίες, η ανάπτυξη λογισμικού ακόμα και σε ένα ε, σύστημα παραγωγής, βιομηχανικής παραγωγής, είναι εργαλεία που είναι διαθέσιμα παντού. Έτσι, αυτές οι διασυνδεδεμένες επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συμπεριλαμβάνονται στην βιομηχανική αλυσίδα εφοδιασμού. Πολύ θεμελιώδου σημασία σε αυτό το στοιχείο και αυτό θα ενισχύσει την ε, ανταγωνιστικότητα, δηλαδή ότι έχουμε επιχειρήσεις που ε, έχουν βαθιές ρίζες στην οικονομία της Ευρώπης και μετά έχουμε και μικρότερες επιχειρήσεις που ε, τροφοδοτούν την επιτυχία αυτών των επιχειρήσεων, των μεγαλύτερων. Αυτό λοιπόν αφορά ζητήματα όπως τα συστήματα πληρωμών, αλλά και ως ε, αφετηρία των καινοτόμων επιχειρήσεων. Γιατί έχουμε και νέους που θέλουν να δημιουργήσουν τέτοιες ε, επιχειρήσεις. Πλούσιο τελικό λοιπόν εδώ. Αυτά από πλευράς μου. Η κυρία Πίτεκαν έχει το λόγο. Και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Καβαρέρο Σάντσες. Ο κύριος Καφεράλτη. Παρακαλώ. Uh, ευχαριστώ πολύ. Πολλά και σημαντικά ήδη υπόθεσαν. Και τα υποστηρίζω στην πλειοψηφία τους. Και εγώ ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά. Θα προσπαθήσω να μην ασκήσω κάποιο κήρυγμα, αλλά είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου αν θέλετε, η οπτική γωνία της βιομηχανίας και ειδικά το θέμα της αποτελεσματικής χρήσης των πόρων. Το μείζον ζήτημα είναι ότι η Ευρώπη θα πρέπει πραγματικά να αναλάβει την επανεκβιομηχάνηση της Ευρώπης. Χρειάζεται λοιπόν μια βιομηχανική δομή, είναι καλό για όλους, για την οικονομία, για τον καταναλωτή, για όλους μας. Από εκεί και πέρα Τίθεται το ερώτημα πώς θα γίνει αυτό. Τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Θέλουμε να ανταγωνιστούμε τις χθεσινές αγορές, τις σημερινές ή ακόμη καλύτερα τις αγορές του αύριο. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς μεγάλος οικολόγος ή να υποστηρίζει ειδικά ε, την αρχή της βιωσιμότητας και σε θήκο επίπεδο για να σκεφτεί ότι θα πρέπει σύντομα να αντιμετωπίσουμε σοβαρά το θέμα της εξάντλησης των πόρων. Άρα πώς θα δημιουργήσουμε τέτοιες αγορές και τέτοια προϊόντα που να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους. Χρειάζεται λοιπόν να παράκουμε τον πλούτο ε, που χρειάζεται οικονομία και η κερδοφορία των επιχειρήσεων αλλά και το όφελος για τους καταναλωτές με μόλις το 10% αυτό που χρησιμοποιήσουμε στο παρελθόν. Χρειαζόμαστε λοιπόν να δούμε το θέμα από την ευρωπαϊκή οπτική του γωνία. Θα πρέπει δηλαδή στρατηγικά να δούμε το θέμα όπως έχουν το το 2020 και άλλες ε, επιμέρους στρατηγικές. Όπως είχαμε μια στρατηγική για το περιβάλλον κτλ. Αντίστοιχη στρατηγική χρειάζεται και εδώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για το μέλλον μας, αλλά και για την επιτυχία της στρατηγικής επανεκβιομηχάνησης, που ελπίζω να διαδραματίσει πολύ σημαντικό και ισχυρό ρόλο στην την έκθεση και ελπίζω η συγχύτρια να δεχτεί προς αυτή την κατεύθυνση κάποιες τροπολογίες που θα υποβάλω. Ο κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα της βιομηχανικής πολιτικής είναι μίζωνος επικαιρότητα στην Ευρώπη για λόγους που μας υπενθύμησε και η Συγχύτρια και η προλαλήσατε συνάδελφοι. Είναι κάτι απόλυτο και ιδιαίτερα σε μια φάση τόσο βαριάς κρίσης όπως αυτή που βιώνουν όλα τα κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν το να φαντάζεται κανείς ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή οικονομία δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς χωρίς μια αντίστοιχη αξία βιομηχανική πολιτική για όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης και ιδίως είναι μια βιομηχανική πολιτική που να συντονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα αναγκαία που θα πρέπει να τα λαμβάνουμε υπόψη κάθε φορά που βλέπουμε αυτό το ζήτημα. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να υπερασπιστούμε με την αναδιάρθρωση ε, όσον ήδη έχουμε, διότι χάνουμε πολλές δραστηριότητες που κατευθύνονται προς υποανάπτυξη χώρες, όπου οι όροι ανταγωνιστικότητας είναι πιο ευνοϊκές για τις επιχειρήσεις, γιατί το κόστος είναι χαμηλότερο και αυτή η διαδικασία επανεκβιομηχάνησης δεν μπορεί να σταματήσει τα σημεία ή στους χώρους που υπάρχει κρίση για να αντιστραφεί ε, η διαδικασία. Θα πρέπει να προσαρμοστεί και το προϊόν και η βιομηχανική διαδικασία. Το πρόβλημα είναι γενικότερο. Η μηχανική πολιτική χρειάζεται την έρευνα και την κοινοτομία σε μεγάλη κλίμακα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε το μέλλον της Ευρώπης χωρίς τα υλικά αγαθά που δημιουργούνται εδώ να παραμένουν αυτά τα παραδοσιακά που θυμόμαστε στο μυαλό μας. Άρα χρειάζεται λοιπόν μεγάλη δουλειά σε επίπεδο έρευνα και καινοτομία εδώ και για το επίπεδο των προϊόντων, τη παραγωγή προϊόντων, αλλά και των παραγωγικών δομών. Το τρίτο θέμα που είναι και αυτό σημαντικό είναι η ολοκλήρωση και η ενίσχυση των μεγάλων ευρωπαϊκών υποδομών, βαρέων και ελαφρών φριών. Μιλάμε για τα οδικά δίκτυα, για σιδηροδρόμους και Δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγική δραστηριότητα που να παράξει πλούτο και άρα να, να ε, ε, ενισχύσει το κεφάλαιο που επενδύεται όταν υπάρχουν ευάλωτες και δύναμες ε, υποδομές. Όταν υπάρχει μια υπερτίμηση της επένδυσης του επιχειρηματία λόγω του κόστου μεταφορών και λόγω της διοχέτευσης ε, των προϊόντων μέσα στον οδών που θα πρέπει να πάρουν, ε, τότε δεν μπορεί αυτή τη διαφορά, αυτή την υπερτίμηση που πληρώνει, να την βρει ε, από πουθενά. Άρα λοιπόν πρέπει να προσαρμοστούν οι υποδομές, οι υποδομές στην Ευρώπη. ιδίω σε ό,τι αφορά την επακινητοποίηση των δραστηριοτήτων που ιστορικά και παραδοσιακά ε, λάβαναν χώρα στην Ευρώπη. Αυτές είναι οι σκέψεις μου που ήθελα πιστεύω να επισημάνω και είναι καλό να σκεφτούμε. Μπορούμε λοιπόν να αναδιοργανώσουμε τη βιομηχανία έρευνα και καινοτομία, το όλο σύστημα της γνώσης, αν θέλετε, είναι πρώτη απόλυτη προτεραιότητα για την πολιτική και ενίσχυση των υποδομών ως ε, στοιχείο της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. Thank you very much. I... Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ ότι το ζήτημα της υποδομής ε, είναι πολύ σημαντικό αλλο κανεί, ε, κύριο Καβελεροσέντης, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε την ευκαιρία να εξηγήσω με δύο λόγια το δικό μας ε, σκεπτικό. όχι μόνο κατά την προετοιμασία της ανακοίνωσης, αλλά και κατά την διάρκεια της υλοποίησής της, γιατί αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Σας ευχαριστώ για τη θετική υποδοχή και τα σχόλια που άκουσα σήμερα εδώ. Υπάρχουν δύο παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω. Αυτή η ανακοίνωση δείχνει ξεκάθαρα ε, τη θέση της Επιτροπής ότι η βιομηχανική πολιτική πρέπει να είναι σπονδυλική στήλη πάνω στην οποία βασίζονται και άλλες πολιτικές ε, έχουμε, περνάμε δύσκολους καιρούς, έχουμε χάσει πάνω από 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ε, στις, ε, στη βιομηχανία τα τελευταία πέντε χρόνια. Και έτσι πρέπει η απάντησή μας να είναι και αντιστοίχως ρεαλιστική. Η ανταγωνιστικότητα είναι μακροπρόθεσμος στόχος και αυτό είναι, συμβαίνει αρκετά χρόνια. Τώρα όμως έχει έρθει η ώρα πράγματι να έχουμε αυτά αποτελέσματα και αυτά να φτάσουν στην αγορά. Για να γίνει αυτό πρέπει να αναλάβουμε δράση. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση, ούτε και κάποιο μέσο κεντρικού σχεδιασμού σε αυτό που έχουμε υποβάλει. Ουσιαστικά έχουμε προτείνει έναν αριθμό τομέων όπου όλοι και όχι μόνο οι Ευρώπη πιστεύουν και σας καλώ να εξετάσετε και τις ε, θέσεις Ομπάμα και του Λευκού Οίκου για τη μηχανική πολιτική, θα δείτε λοιπόν ότι εδώ έχουμε εντοπίσει κάποιους τομείς, όχι για την επιλογή νικητών, αλλά ως τομείς που θα, θα αναπτύσσονται ε, ταχύτερα στο βραχυπρόθεσμο μέλλον. Και δεύτερον, θεωρούμε ότι αν ε, θέσουμε αυτά τα μέσα στη διάθεση Τη Ευρωπαϊκή οικονομία, σε ό,τι αφορά την αγορά ε, και επενδυτικά μέσα, θα έχουμε τα κατάλληλα αποτελέσματα. Έχουμε επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε αυτά τα ζητήματα. Τα, προγράμματα πλαίσια για την ανάπτυξη και την, ε, για την έρευνα και ανάπτυξη τρέχουν εδώ και χρόνια και ε, δυστυχώς σε πολλά από αυτά τα προγράμματα τα στοιχεία έρευνας και ανάπτυξης, τα βραβεία Νομπέλ μας και το καθεξής δεν τα έχουμε μεταφράσει ε, σε βιομηχανική αριστεία και στον ηγετικό μας ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες στην αγορά, προκειμένου να αναπτυχθούν αυτές οι αγορές. Υπάρχουν ορισμένες τις αγορές που είναι έτοιμες να αναπτυχθούν. Για παράδειγμα, στα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Ε, σίγουρα θα αναπτυχθούν στο μέλλον και το ξέρουμε. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε τις επενδύσεις ε, για όλες τις υποδομές σε ό,τι αφορά αυτές τις υποδομές που θα πρέπει να διαμορφωθούν για να υποδειχθούν αυτή τη νέα γενιά αυτοκινήτων. Δυστυχώ υπάρχουν ε, δύο πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί ιδιωτικά στην Ευρώπη και παρά τις συστάσεις της Ευρώπης, της Επιτροπής, η βιομηχανία δεν έχει συμφωνήσει. Και αυτό κρατά πίσω αυτές τις ε, επενδύσεις. Και δεν μπορούμε να μένουμε πλέον με σταυρωμένα τα χέρια. Θα μπορούσα να αναφέρω κάποια παραδείγματα στις βιοτεχνολογίες, σε πολλούς τεχνολογικούς τομείς. Ε, επιστημονική γνώση υπάρχει που είναι έτοιμη να υλοποιηθεί αρκεί να ε, διαμορφώσουμε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να εμπιστευτούν μία την άλλη και να συλλέξουν αυτά τα ε, στοιχεία τεχνολογίας που είναι τα κομμάτια του πάζελ. Γενικά θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε αυτά τα βήματα διαμορφώνοντας αυτές τις συνθήκες και μετά στο τέλος θα δούμε αν, ότι θα υπάρχει μεγάλη... Αν θα υπάρχει, αν αυτή η μεγάλη ανάπτυξη θα υπάρχει στις βιοτεχνολογίες ε, ή στα αυτοκίνητα. Αυτό θα το δούμε. Όμως οι επιχειρήσεις ε, θα πρέπει να δράξουν ε, αυτές τις ευκαιρίες. Και αυτές θα αποφασίσουν. Υπάρχει μια έκθεση McKenzie του τελευταίου Δεκεμβρίου. Σας καλώ να τη διαβάσετε και εκτιμά ότι οι ιδιωτικέ επενδύσει ε, στην Ευρώπη έχει πέσει κατά 350 δι από την 2007 μέχρι το 2011. Το 2011, στο τέλος αυτής της περίοδου, υπήρχαν 750 δισεκατομμύρια ευρώ που κάθονταν ουσιαστικά στους ισολογισμούς ε, των 100 μεγαλύτερων επιχειρήσεων ε, της Ευρώπης. Υπάρχει λοιπόν η ρευστότητα που απαιτείται για αυτές τις επενδύσεις και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα μηνύματα που μεταβιβάζουμε στην, ε, στις επιχειρήσεις για να είμαστε σίγουροι ότι θα διαμορφωθεί το κατάλληλο ε, περιβάλλον για να ξεκινήσει νέα ροή κεφαλαίων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ανάπτυξης. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας αλλά και για την παραπομπή σας στην Επιτροπή Μακέντζη. Ευελίν, μας έχει δώσει ήδη το χρονοδιάγραμμα, κάποιε καταληκτικές πληροφορίε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εδώ παρόντες για την ε, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που μου έδωσε ε, τροφή για σκέψη. Αλλά θα απευθύνω για άλλη μια φορά ε, το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να επισημάνω ότι φαίνεται να έχει κάνει πολύ καλή δουλειά το λόμπι της βιοτεχνολογίας στην Επιτροπή, γιατί όπου και να ειστρέψω το βλέμμα, οποιοδήποτε θέμα και να με απασχολεί που σχετίζεται έστω και ε, μακρόθεν με το θέμα αυτό της βιοτεχνολογίας, πάντα το βλέπω να εμφανίζεται στις συζητήσεις. Και αυτό που με ανησυχεί είναι ακριβώς σε σχέση με τη λεγόμενη προγραμματισμένη οικονομία, σχεδιασμένη οικονομία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, αυτό που εξήγησα και επιμένω ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε επακριβώς από πού ακριβώ οι τεχνολογιακές. Θα συμφωνήσω αυτό που είπατε ότι χρειάζονται και οι συνθήκες πλαισίου ώστε να αφήσουμε ε, ε, πεδίο ελεύθερο στη δημιουργικότητα. Μην προσπαθούμε εκεί που ήδη έχει γίνει κάτι και εκεί που προσπαθούν και εκεί που έχουν κάθε δυνατότητα για να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις να δώσουμε υποστήριξη. Γιατί να βοηθήσουμε αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνολογία, να βοηθήσουμε τους λεγόμενους startups, αυτούς που τώρα αρχίζουν τις προσπάθειές τους. Σε αυτό θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στραφεί και να κοιτάξει τι κατεύθυνση θα επιλέξει. Πάντως η κατεύθυνση που επιλέγει δεν με βρίσκει σύμφωνη μέχρι τώρα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Πολλές σωστές εύστοχες παρατηρήσεις ακούστηκαν βελτίωση της αγοράς των ε, εμπορικών προϊόντων. Κύριε Σφάπ, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Το διαδικό σύστημα στην ε, απόκτηση δεξιοτήτων, ε, μόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση στη Γερμανία έχει δώσει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και από την χώρα της πρώτης μου καταγωγής ξέρω ότι υπάρχει θεωρητική γνώση σε υψηλό επίπεδο στην νεολαία, αλλά όχι πρακτική. Και γι' αυτό δεν μπορούν να υλοποιήσουν, να θέσουν σε εφαρμογή αυτά που ξέρουν. Και σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σα για τι ε, τράπεζε βιομηχανική ανάπτυξη, κυρία Χατζημαρκάκη, βεβαίω να το συζητήσουμε. Είναι ενδιαφέρον. Καθυστερήσει στι πληρωμορομέ και εκτέλεση. Βεβαίω, αλλά, αλλά μήπω εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποιο ζήτημα εσωτερική πολιτική τη Γερμανία, κυρία Χατζημαρκάκη. Ή να το πω διαφορετικά. Γιατί η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας δεν αξιοποιεί την ε, οδηγία για την υπερημερία στις πληρωμές που είναι μια ε, οδηγία ελάχιστης εναρμόνισης ώστε να ρυθμίσει το ζήτημα και στη Γερμανία ένα ζήτημα και ένα πρόβλημα που χρονίζει. Ε, περιμένω να γίνει ο κύριος Χατζημαρκάκης υπουργός Οικονομικών για να το συζητήσουμε. Για το ισχυρισμένη οικονομία. Κυρία ρουλέφη. Εν πάση περιπτώσει. Ο σχεδιασμός μάλλον των πόρων ε, είναι ασφαλώς μια καλή ιδέα, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ε, περιλάβουμε στις προτάσεις. Να ορίσουμε δηλαδή στόχους, να λέμε τι θέλουμε. Θέλουμε αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση των πόρων, θέλουμε αποτελεσματικότητα στη χρήση της ενέργειας, όλα αυτά τα πράγματα τα εντάσσονται εν τέλει στην βιομηχανική πολιτική, ώστε η έρευνα και η επιστήμη να στηριχθούν, γιατί και χρειαζόμαστε χρήματα, με αποτέλεσμα να αφήνουμε ελευθερία στις ε, επιχειρήσεις να επιλέγουν αυτό που θέλουν, αλλά ταυτόχρονα και την επιλογή στον πολίτη για το τι είδους ενέργεια ε, προτιμάει, να μην τα ορίζει αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτός είναι ο σωστός τρόπος, ασφαλώς θα το προτείνω και ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Και ευχαριστώ και εσάς κύριε Χάρμπορ βεβαίως για, για τις δικές σας παρατηρήσεις, για την ε, ε, οικονομία με τις οποίες συμφωνώ επίσης. Για τον κύριο Σουάπ επίσης είπατε ότι δεν συμφωνείτε με τον ελάχιστο μισθό στο σημείο 4. Μα εγώ δεν έχω βάλει τέτοια παρατήρηση. Δεν το έχω καταγράψει αυτό. Ανέφερα ότι έχω αυτή την ιδέα. Γιατί εγώ, αν κοιτάξει το κείμενο, δεν μιλάω για ελάχιστο μισθό. Και επίση. Πιστεύω ότι θα πρέπει η συζήτηση να μην περιοριστεί σε αυστηρούς όρους ποιος έχει πια αναρμοδιότητα. Εάν θέλουμε να δώσουμε λύσεις που θα βοηθήσουν την ιστορική αγορά θα αγγίξουμε και θέματα της βιομηχανικής πολιτικής. Έχουμε δικαίωμα να τοποθετηθούμε και εγώ την πρόταση αυτή θα την καταθέσω έστω και αν δεν είστε σύμφωνος. Πάντως περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση. Good. Well, it's been an excellent debate. Εξαιρετική αυτή η συζήτηση. Είναι Μια συζήτηση που θα πρέπει να επαναλαμβάνεται πιο συχνά. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή τους. Κατανοούμε πως και την απουσία κάποιων γιατί υπάρχει και έργο που τρέχει σε άλλες επιτροπές. Ξέρω ότι θα έχουμε και πολύ των εισήτησεων που θα λάβουμε και πολύ ενδιαφέρουσε τροπολογίες. Ας περάσουμε τώρα σε δύο πολύ ε, σημαντικές γνωμοδοτήσεις που εκπονούμε ενώ κύριε Αρμόδια Επιτροπή Νιεκών δεν υπάρχει ακόμη επίσημη αίτηση για ενισχυμένη συνεργασία. Πιστεύω ότι αυτή η πρόταση θα απορριφθεί, διότι δεν έχουμε καταφέρει τελικά να περάσουμε τη θέση μας. Το ίδιο κάναμε και σε άλλες περιπτώσεις, ιδίως στην περίπτωση του ιατρικού ε, εξοπλισμού τρικών που ήταν πραγματικά πολύ ατυχές. Αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει απλά να υποβάλουμε τροπολογίες και να ελπίζουμε να γίνουν αποδεκτές από την αρμόδια επιτροπή. Και ο εισηγητής θα μας πάρει στα σοβαρά, γιατί θα τους έχουμε πλημμυρίσει με τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα, θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση για τα έγγραφα μαζικές πληροφορίε σχετικά με επενδυτικά προϊόντα, με εισηγητή τον κύριο Πιεραντώνιο Παντσέρη. Είναι εδώ κυρία Ρούλερ για τους Πρασίνους και άλλοι συνάδελφοι για όλες τις ομάδες και την ομάδα μου ανεπισήμως είμαι ο Σκιώδης. Δεν έχουμε βάλει τροπολογίες και έχουμε και πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι δεν είναι. Είναι κανείς εδώ. Πάντως δεν είναι στα χαρτιά μου. Θα δώσουμε πάντως το λόγο στην Κομισιόν να δούμε ποιος είναι εδώ εκ μέρους της Επιτροπής για να τον ανακοινώσουμε. κύριος Λούτε εξ ονόμας Επιτροπής. Ναι, ωραία. Λούτε, καλά λέω το όνομά σας. Ωραία. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν είναι πολύ καλές οι σημειώσεις μου, οπότε θα σου δώσω το λόγο αργότερα. Ο κύριος Παντσέρη, παρακαλώ αν θέλει να μας μιλήσει για τις τροπολογίες. Θέλετε να κάνετε κάποιο ερώτημα. Αν κατάλαβα καλά η ΕΚΟΝ και για το MT2 καθυστερήσε την αρχική συζήτηση για τις 27 Μαΐου. Άρα έχουμε πιο πολύ χρόνο για το θέμα αρμοδιότητας. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να το διευκρινίσουμε διότι η Επιτροπή μας έχει πολύ καλύτερη εξουσία επί του θέματος από ότι αυτή τη στιγμή. Αν έχω καταλάβει σε θέματα προστασίας καταναλωτή και δικαιώματα του καταναλωτή, είναι πολύ διαφορετική προσέγγιση της εικόνα από τη δική μας. Αν ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα, καταφέρουμε στη σωστή ισορροπία, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι σημαντικό για θέματα καταναλωτή. Το θέμα λοιπόν της αρμοδιότητας είναι σημαντικό επειδή αποτύχαμε στο παρελθόν, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε στο μέλλον. Ναι, μα το προωθήσαμε το θέμα όσο μπορούσαμε. Πήγε μέχρι τη διάσκεψη των Προέδρων το θέμα και εν μέρει το πρόβλημα είναι ότι η ΕΚΟΝ δεν θέλει να μπει σε καμία ουσιαστική συζήτηση από του θέματο. Απλά μας απαιτώνει μια επιστολή που μα απορρίπτει όλα τα αιτήματα, άρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Και εγώ έτσι απλά δεν μπορώ να ζητώ συνεδριάσεις. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Από την άλλη, γνώμη μου είναι, αν η δική μας ψηφοφορία ορίζεται αρκετά νωρίτερα από τη μέθοδο εργασίας που ακολουθεί ΕΚΟΝ, τότε έχουν πιθανότητες να περάσουμε τα βασικά μας μηνύματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Θα πρέπει να δουλέψετε σκληρά στους συζητητές για να περάσει την άποψή σας. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό θέμα η προστασία του καταναλωτή. Δεν θα πρέπει λοιπόν να καθυστερούν προσφορές ιδίω στη δική σας έκθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικό εμεί να έχουμε τελειώσει το θέμα αυτό όταν θα ξεκινήσει να το συζητά η εικόνα. Η Εύελιν θέλει το λόγο. Είπατε μόλις, Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να αποφασίσει ακόμη η διάσκεψη των Πρόεδρων. Άρα δεν έχει ληφθεί ακόμα αποφασή επίσημη. Γι' αυτό θα πρότεινα να περιμένουμε, αφού η αρμόδια καθήλυν επιτροπή φαίνεται να αναβάλει τη λήψη αποφάσεως, ας καθυστερήσουμε κι εμείς. και θα πρότεινα να αρχίσει τη δουλειά ο εισηγητής με τους και εισηγητές σαν να ήμασταν συναρμόδια ή αρμόδια για γνωμοδότηση επιτροπή και μετά αναλόγως της αποφάσεως να δούμε και να πράξουμε. Γιατί όσο δεν υπάρχει επίσημη υπόθεση δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε πιο πολλές προσπάθειες και να πιεστούμε περισσότερο. Είναι κάτι πάντως πρέπει να συζητήσουμε και με τους επικεφαλείς των πολιτικών μας ομάδων, γιατί εγώ βλέπω ότι είναι λυπηρός ο τρόπος με τον οποίο σε τόσο σημαντικούς τομείς ξεσπάνε ε, αντιπαραθέσεις πολιτικού χαρακτήρα. Και βλέπω ότι ε, τον τελευταίο χρόνο τελικά χάσαμε τόσα πολλά όλοι σε τομείς που είχαμε αρμοδιότητες ή συναρμοδιότητα έστω, λόγω της απόρριψη πλευράς του Προέδρου της Διασκέψης των Προέδρων, του κύριου Λένα, μιας πρότασης. Γι' αυτό καλό θα ήταν να κοιτάξουμε πόσοι, πόσες εξουσίες μπορεί να έχει ένας βουλευτής, μεμονωμένος βουλευτής, έστω και πρόεδρος της Διάσκεψης των Πρόεδρων, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Εγώ θεωρώ απαράδεκτο να χάνει η Επιτροπή μας διαρκώς αρμοδιότητες. Δεν γίνεται. Δεν επιτρέπεται. Λοιπόν, το θέμα αυτό θα επανέλθει το απόγευμα στους συντονιστές. Υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις για το χρονοδιάγραμμα. Ε, ε, εξαρτώμεθα βεβαίως από τους εισηγητές επί του θέματος. Το τι θα κάνουμε τελικά στο θέμα της αρμοδιότητας μεταξύ των επιτροπών, αυτό θα είναι αντικείμενο της συζήτησης που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Οπότε όλα αυτά που είπατε θα ανακύψουν συζήτηση, διότι πράγματι η όλη δικασία αυτή τη στιγμή δεν είναι απόλυτα διαφωνία. Κύριε Σουάμ, θέλετε το λόγο. Πολύ σύντομο για το ΕΛΚ και το λέω και εξ τη κυρία Σπιτκάνιν που είναι η σκιώδη. Η καθυστέρηση δεν είναι πρόβλημα. Αν δείτε όμω την ουσία και τη σύγκρουση αρμοδιοτήτων και στην περίπτωση της ε, έκθεσης Μπερές, Εκεί είχαμε τα μεγαλύτερα προβλήματα με την Επιτροπή μας και θέλουμε να συνομιλήσετε με την κυρία Περές πριν τη συζήτηση που έχετε με τους άλλους πρόεδρους των Επιτροπών γιατί εκεί είχαμε την πηγή του σημαντικότερου προβλήματος που ξεκίνησε τους τελευταίους αυτούς μήνες. Ναι, πράγματι οι εισηγητέ δεν ε, είναι πάντα τόσο πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί μα. Εντάξει, α το θέσουμε έτσι. Προχωρούμε. Από πρακτική πλευρά συμφωνώ απολύτω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε, στους τομείς της προστασίας καταναλωτών ε, που υπάρχει ζήτηση για ενισχυμένη συνεργασία. Δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξουμε αυτό. Πρέπει να φροντίσουμε και να εργαστούμε επιμελώς. Ο Κύριε Παντζέρη, θέλετε να δώσετε τη γνώμη σας για τις ε, τροπολογίες και μετά να δώσετε το λόγο στους Χιώδης. Κύριος Παντζέρη. Ευχαριστώ. Εννοείται ότι και εγώ συμφωνώ. Πρέπει να βρούμε μια αίσια έκβαση για, αυτή την, για αυτό το πρόβλημα και αυτή τη σύγκρουση, γιατί δεν μπορεί τελικά οι αποφάσει που λαμβάνονται από μια άλλη επιτροπή του Κοινοβουλίου να λειτουργούν ει βάρο των καταναλωτών. Πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Σε κάθε περίπτωση, να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις για τη δουλειά που έγινε ως τώρα και ιδίως για τις σκέψεις που εξέφρασαν και στη χθεσινή συνεδρίαση που οργανώσαμε χθε για να συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. 16 συμβαστικές τροπολογίες που εστιάζουν κυρίως στη μορφή ε, και το περιεχόμενο, άρθρα 6, 8 και 11 και το μηχανισμό εναλλακτική επίλυση διαφορών, άρθρο 15. Πολλές από τις τροπολογίες ε, έτυχαν ευρεία συνένεσης, όπως για παράδειγμα η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή, ο αποκλεισμός αναφοράς σε ε, ε, διαφημιστικά μηνύματα, η αναφορά στους εκπρόσωπους κινδύνους που συνδέονται με το προϊόν και αυτούς που αφορούν και τον ενδιάμεσο, και έπειτα υπάρχει μια πρόταση. Θεωρούμε ότι η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνοδεύεται από ε, την ε, τεχνική πυροχνομοσύνη των αρμόδιων φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για την ελεκτική επίλυση διαφορών. Πολλές τροπολογίες ε, υπέβαλα, όσο στο διατακτικό να έχουμε και καλύτερη εξήγηση αυτού του τρόπου επίλυση διαφορών. Και αναφέρομαι επίση και στην ευθύνη των κρατών μελών να εγγυηθούν την ορθή διεξαγωγή ε, της όλης διαδικασία ώστε να υπάρχει καλή ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με δυνατότητα χρήση αυτή τη λύση, όπω και δυνατότητα και ομαδική συλλογική επίλυση διαφορών. Οι άλλε σκιώδει πρότειναν να γίνει παραπομπή στην οδηγία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Επ' αυτού και για άλλα τεχνικά ζητήματα που δεν υπάρχουν διαφορετικά απόψεις, όπως το σύστημα ταξινόμησης και για το εύρος του κειμένου και το άρθρο 8.5, το επόμενο διάστημα θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε και σε άλλες τροπολογίες για να υπάρχει και μέγιστη δυνατή συνένεση. Κατά λοιπά, λαμβάνοντας υπόψη για την οικότερη θέση των σκιωδών και το θετικό επικοδομητικό ε, κλίμα, πιστεύω ότι σύντομα θα καταλήξουμε σε μία κοινή θέση πριν την ψηφοφορία στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Uh, well, thank Σας ευχαριστώ για τη εργασίες σας με τους ε, σκιώδεις, ε, για την επίτευξη των συμβαστικών Κυρία Πιδγάινεν, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή για την εξαιρετικά γόνιμη συνεργασία. Πριν περάσω στην ίδια την έκθεση, να αναφερθώ και στο ζήτημα της συνεργασίας με τις ε, υπόλοιπες επιτροπές. Και πράγματι, η κατανάλωση, η προστασία των καταναλωτών αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Όχι μόνο για τα οικονομικά ζητήματα, αλλά και για τη μεταφορά και τα δικαιώματα των επιβατών. Πολύ ουσιαστικά. Τώρα, για αυτή την νομοθεσία, ελάβαμε το κείμενο των συμβαστικών χθες είχαμε μια γενική συζήτηση επί της αρχής και ακόμα εξετάζουμε τις διατυπώσεις, στο ίδιο το κείμενο, αλλά φαίνεται ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, από πλευράς μας, το ζήτημα του πεδίου εφαρμογή έχει συζητηθεί επί μακρόν. Είναι προς όφελος του καταναλωτή ε, και των ίσων ορών ανταγωνισμού, το πεδίο εφαρμογή να, εφαρμογής να διευρυνθεί για να συμπεριλαμβάνει διαφόρων ειδών ε, προϊόντων. Με την εξαίρεση βέβαια κάποιων ομολόγων και λογαριασμών. Όμως πρέπει να δούμε πόσο ακριβώς θα χειριστούμε το ζήτημα, γιατί η κατάσταση Πρέπει όμως να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και με την Επιτροπή. Δεύτερο στοιχείο, όπου είχαμε θετικά αποτελέσματα, είναι οι διάφοροι τύποι καταναλωτών. Και εγώ και η μητέρα μου, για παράδειγμα, είμαστε καταναλώτριες, με διαφορετικές ανάγκες όμως και πληροφόρησης. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει αυτή η εργαλειοθήκη που να είναι αρκετά ευέλικτη για διάφορα είδη καταναλωτών. Τώρα, για την έκταση του ε, εγγράφου και για να είναι ώστε να τον πιο σαφές, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τις δαπάνες και πιο ξεκάθαρες διατυπώσεις, ούτως ώστε οι καταναλωτές που χρειάζονται αυτές τις ε, ευανάγνωστες και εύληπτες ε, πληροφορίες να τις έχουν και πρέπει να υπάρχει και παραπομπή σε άλλα κείμενα, γιατί ίσως κάποιοι καταναλωτές να θέλουν λεπτομερέστερες πληροφορίες για το προϊόν. Μετά αυτό συνδέεται βεβαίως και με τον ε, κίνδυνο. Ο καταναλωτής κατανοεί τον κίνδυνο. και εφόσον τον κατανοεί μπορεί να αποφασίσει να αποφασίσει αν ε, θέλει να αναλάβει αυτό τον κίνδυνο ή όχι. Δεν είναι πάντα κακός βέβαια, κακό αυτό το ρίσκο. Γιατί το ρίσκο πολύ συχνά συνδέεται και με το, με, με το έπαθλο, Και αυτό συνδέεται και με τη δομή των δαπανών ή του κόστους, γιατί και αυτό μπορεί να αποτελέσει ρίσκο για τον επενδυτή. Αν κάποιος είναι σίγουρος ότι σε αυτές τις δαπάνες με αυτές τις δαπάνες δεν μπορεί κάποιος να ε, αντισταθμίσει τον πληθωρισμό ή μπορεί μάλιστα να βρεθεί και να μπει και μέσα όπως λέμε, τότε μπορεί απλά να βάλει τα χρήματά του σε ένα καταθετικό λογαριασμό. Γι' αυτό και η δομή των δαπανών και ε, ο σωρευτικός αντίτυπος αυτών θα πρέπει να είναι και πάλι ε, στοιχεία εύληπτα για τον καταναλωτή και έτσι γλιτώνουμε κάποιες από αυτές τις παγίδες που βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο σε τέτοιου είδους επενδύσεις. Μετά, σε ό,τι αφορά το παρελθόν ή το μέλλον, ε, σε ό,τι αφορά τις ε, επενδυτικές επιλογές. Γενικά υπάρχουν ισχυρά κίνητρα για να υπάρχουν ε, επιχάρτω αυτές οι αναπτυξιακές στρατηγικές μαζί με τα διάφορα σενάρια, συμπεριλαμβανομένου και, του, και της χειρότερης ε, περίπτωσης. Τέλος, πώς επιλύονται οι διαφορές και εδώ υπάρχει η αναφορά στα συστήματα EDR και είναι καλό να υπάρχει δισταυρούμενη παραπομπή με την ομοθεσία και εδώ. Και μετά υπάρχουν κάποια διευκρινιστικά στοιχεία και παραπομπές ε, στη διαφήμιση. Θα πρέπει να αναφέρονται αυτά, αλλά δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε. Ευχαριστώ. Um, ευχαριστώ, κύριε Σόι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ δεν ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτό το θέμα. Η γνωμοδότησή του είναι πολύ καλή βάση για συζήτηση και η συμβαστική του και οι συμβαστικέ τροπολογίες δείχνουν αυτό. Γενικά, έχουμε να κάνουμε ένα ακριβές και εύληπτο μη παραπληκτικό κείμενο. Πρέπει να είναι επίσης ένα εργαλείο που να διευκολύνει την συγκρισιμότητα μεταξύ των επενδυτικών προϊόντων της αγοράς. Θεωρώ ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια ευέλικτη προσέγγιση. Λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλιών και Συντάξεων και την ε, αρμοδιότητα που έχουν για την ανάπτυξη ρυθμιστικών προτύπων σχετικά με αυτές τις πληροφορίες. Στο προσεχηματικό σημείωμα αναφέρεται ρητός ότι το kit δεν είναι μία σύσταση για την αγορά του προϊόντος και ούτε είναι εξαιρετικό, Δηλαδή, ο μικροεπενδυτής καλό είναι να διαβάσει και άλλα στοιχεία πριν αποφασίσει. Το κόστος, ευαίσθητο και σημαντικό ζήτημα. Θα πρέπει ο καταναλωτής να πληροφορείται για το κόστος. Γιατί αυτό σίγουρα επηρεάζει την απόδοση επί της επένδυσης. Έπειτα, πληροφορίες για το φορολογικό καθεστώς είναι χρήσιμες. Δεν είναι εύκολο πάντοτε να δίνονται αυτές τις πληροφορίες, ιδίως όταν είναι ηλεκτρονική η αγορά. Όταν όμως είναι δυνατόν να υπάρχουν και αυτές οι πληροφορίες. Έπειτα, οι μικροί επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν κατά πόσο υπάρχουν και όροι, προϋποθέσεις στην αγορά δηλαδή κατά πόσο χρειάζεται να κάνουμε μια ελάχιστη αρχική επένδυση ή όχι. Σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα του προϊόντος. Και εδώ επέβαλα κάποιες σχετικές τροπολογίες, όπως και άλλοι συνάδελφοι. Θα πρέπει να προειδοποιούμε τους επενδυτές ότι η παρελθούσα απόδοση δεν είναι α, εγγύηση απόλυτη για τη μελλοντική απόδοση. Και ο κ ότι το τι θα πρέπει να δίνει πληροφορίε τέτοιε ώστε ο μικροπαιδευτή να μπορεί να συγκρίνει την απόδοση του προϊόντος, του πολιτικού προϊόντος με κάποια benchmarks. Από και πέρα με τον κατάλογο βλέπω πολύ αρνητικά το ενδεχόμενο αρνητικών α, στοιχείων στο σύστημα. Αξιοπιστία τώρα των επενδυτικών προϊόντων θα πρέπει να υπάρχει σχέση αιτίωτια του ανάμεσα στο προϊόν επένδυση και το kit. Ιδάλλως, εκθέτουμε τους ε, κατασκευαστές, τους, ε, ε παρόχους αυτών των μελετικών προϊόντων με ε, υπερβολική ευθύνη. Τώρα, λίγα λόγια για τις αναλλακτικές επιλύσεις διαφορών, το ADR. Το άρθρο της Κομισιόν δεν είναι κατοπλών ευτυχές, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι πρόσφατα συμφωνήσαμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Μαρτίου το πακέτο ADR-ODR. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Δεν μπορούμε λοιπόν εδώ να ξαναλέμε όλα όσα λέει η σχετική οδηγία. Μια απλή παραπομπή θα ήταν καλύτερη. Ιδίως ό,τι αφορά την διαθεσιμότητα ε, εξοδικαστικών μέσων επίλυσης διαφορών. και την αναφορά στο κατά πόσον προσφέρουν αυτές τις δυνατότητες οι ίδιοι ε, οι πάροχοι, οι δημοσιολαβητές. Αλλά και πάλι ε, το σχετικό μέρος του κειμένου δεν είναι σαφές. Μιλάει για το δικαίωμα προσφυγής ένδικα μέσα. Καμία αναφορά δεν γίνεται όμως στις περιόδους παραγραφής ε, και το πώς έρχεται αυτό με την διαφύλαξη του δικαιώματος πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Uh, thank you um, Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ρούλα. Πολύ σύντομα. Δυστυχώς ε, δεν μπορούσα να συμμετάσχω στην ε, συνάντηση των σχεδόν χθε, όμως μεταξύ, έχω δει ότι οι συμβαστικές προτάσεις ε, του κυρίου Παντσέρη είναι πολύ καλέ. τις διάβασα προσεκτικά, σίγουρα θα τις στηρίξουμε. Και τον ευχαριστώ πολύ. Τόμας Ένω. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να είμαι σαφής. Η πρόταση της Επιτροπής για περισσότερη διαφάνεια σε αυτό τον τομέα είναι κάτι που στηρίζουμε. Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις η Επιτροπή δεν πάει, δεν προχωράει όσο θα έπρεπε. Το έγγραφο που συνδέεται με τα λεγόμενα ε, πακέτα προϊόντων δεν είναι αρκετά φιλόδοξο και δεν θεωρούμε ότι ε, οι διευθετήσεις για τις ενστάσεις ή για τα αρνητικά θα πρέπει να εξαιρεθούν. Διότι δεν υπάρχει επαρκής προστασία για τους μικρούς επενδυτές στην πρόταση της Επιτροπής. Οι συμβαστικέ ε, του εισηγητή είναι σωστές και εν γέννη τις στηρίζουμε. Ο κύριος Παντζέρη μιλά για ανεπαρκές ε, πεδίο εφαρμογή τη οδηγία και θεωρεί ότι το, οι δαπάνε για τον μέσο επιχειρηματία επενδυτή θα πρέπει να προσθεθούν για τις δαπάνες που αναφέρει η Επιτροπή. Οι πληροφορίες για τέτοιου είδου δαπάνες θα πρέπει να συμπεριληφθούν Όταν φτάνουμε στην υπόθεση των πληροφοριών που συνοδεύουν αυτό το πακέτο, βλέπουμε μια σύγκριση με τα φαρμακευτικά προϊόντα. Υπάρχει ένα τυποποιημένο ε, συνοδευτικό έγγραφο για οποιοδήποτε φαρμακευτικό προϊόν αυτή τη στιγμή που αναφέρει τους κινδύνους και τον τρόπο χρήσης και δεν βλέπουμε γιατί δεν μπορεί να, χρησιμοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός και στα επενδυτικά προϊόντα. Αν θέλουμε κάτι να είναι συγκρίσιμο και απλό, αυτό πρέπει να κάνουμε. Θέλουμε λοιπόν ένα σύντομο σαφές ε, φυλάδιο στην κατάλληλη γλώσσα. Γιατί δεν μπορεί κανένας βεβαίως να αγοράσει ένα φάρμακο όπου ο φαρμακοποιός είχε την επιλογή να προσθέσει επιπλέον πληροφορίες στο πακέτο ή όχι στη συσκευασία. Δηλαδή δεν είναι ο πολιτής αυτός που έχει την ευθύνη ε, για τις πληροφορίες που παρέχονται με το προϊόν. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος της ε, συμπερίληψης ε, διαφημίσεων εδώ στην πράξη. Τα επενδυτικά προϊόντα οι πολιτές επιθετικών προϊόντων έχουν πλέον την φήμη της ε, μη σωστής παρουσίασης των κινδύνων. Άλλη πρόταση που κάνει ο εισηγητής είναι ότι ο πολιτής θα έχει αρνητικό στοιχείο, θα έχει ευθύνη όπως ακριβώς και το ιατρικό προσωπικό, όπως ο φαρμακοποιός ή ο ιατρό έχουν ευθύνη να πούν στον καταναλωτή ποιο είναι το κατάλληλο φαρμακευτικό προϊόν για εκείνον. Προφανώς όμως και εκείνοι είναι ε, που αποφασίζουν ποιο είναι το κατάλληλο προϊόν. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και με τα επενδυτικά προϊόντα. Να μην έχουμε δηλαδή μόνο τις βασικές πληροφορίες σε αυτό το φυλάδιο, αλλά κάτι παραπάνω. Και τέλος, το βάρος της απόδειξης σε ζητήματα ευθύνης θα πρέπει να ε, το επομίζονται όσοι παρήχαν λαθασμένες πληροφορίες, γιατί κάποιες φορές περιπλέκονται τα πράγματα για τον ε, μικρότερο φορέα. Έτσι, αυτός που έχει παράσει αυτές τις λαθασμένες πληροφορίες, ο εκδότης του φυλαδίου ίσως θα πρέπει να είναι αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη. Αυτές τις ε, προτάσεις μπορούμε να τις στηρίξουμε. Ο εισηγητής ε, έκανε μια πολύ καλή δουλειά. Τον ευχαριστώ και ελπίζω να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στο τέλος. Ωραία, ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και τους κοιότης. Υπάρχει κάτι άλλο. Τότε να δώσω το λόγο στον κύριο Λέντεν, να πει δύο λόγια πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο. Thanks, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. σας ευχαριστούμε για τα σχόλια και τη θετική προσέγγιση της Επιτροπής σας. Είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε τα στοιχεία που αφορούν τους καταναλωτές στα πλαίσια της πρότασης αυτής. Όταν σχεδιάσαμε αυτό το kit, λέμε ναι, θα πρέπει να είναι ένα σύντομο έγγραφο, να χρησιμοποιείτε την κατάλληλη χρονική στιγμή σε συγκεκριμένη και απλή γλώσσα προετοιμάσω την πρόταση. Εξετάσαμε και εμεί θέλουμε πιο πολλέ πληροφορίε, ενδελεχεί πληροφορίε όλου του τομεί ή να έχουμε ένα σύντομο, ένα ευσύνοπτο κείμενο. Και εκεί προσπαθήσαμε να βρούμε μια ισορροπία. Μελετήσαμε με μεγάλη προσοχή τι προτάσει και με χαρά να δούμε κάποια επιμέρου στοιχεία για το τι θα πρέπει να περιλαμβάνει αυτό το kit. Η οδηγία πρίψη είναι επισηματική μαζί με την οδηγία για τις πωλήσει και με τη MIFID και με την οδηγία για τις ασφαλίσεις. Άρα όλες αυτές οι οδηγίες συνδέονται σε κάποια σημεία, σε θέματα δηλαδή πληροφόρησης. Τα θέματα των κυρώσεων και των εναλλακτικών ε, εναλλακτική επίλυση διαφορών. Εκεί παρακολουθούμε τις εξέλιξεις, ε, την αναμοθεσία Κατά την εκπόνηση αυτής της πρότασης βασιστήκαμε στην κείμενη νομοθεσία. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει ε, εγκάρσια, αν θέλετε, συμμόρφωση μέσα στο κεκτημένο. Τώρα, για κάποια ζητήματα τα κατανοούμε ότι για παράδειγμα, η αποδοτικότητα ε, ενός προϊόντος στο παρελθόν δεν είναι εγγύηση και το μέλλον. Το γνωρίζουμε αυτό. Θέλουμε να βρούμε μια καλύτερη διατύπωση και με τη βοηθεία σας. Τώρα, για το θέμα ε, της ύπαρξης ενός φαναριού ή όχι. Το συζητήσαμε αυτό και άλλες περιπτώσεις και λέγαμε ότι μάλλον δεν πρέπει να είναι φανάρι αυτό που να ανάβει ή όχι, αλλά μάλλον μια ε, ζυγαριά που θα κρίνει. Κατά λοιπά, θα απελευθερώσουμε προσοχή της τροπολογίας σας και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Πατσαρή, θέλετε να πείτε κάτι παραπάνω. Ας αφήσουμε το χρονοδιάγραμμα ανοιχτό αυτή τη στιγμή, ανάλογα από το πώς θα εξελιχθούν οι συζητήσεις, ώστε αν κρυθεί αναγκαίο να το στήσουμε το θέμα και πάλι. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για όλες τις τοποθετήσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο-τρία σημεία μόνο. Το πρώτο, για το πεδίο εφαρμογής. Στη συζήτηση που είχαμε εδώ, οι συνάδελφοι τοποθετήθηκαν υπέρ της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής. Είναι σημαντικό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εντάξει αυτή την έννοια Εφή εξ αρχή καθώς είναι η βασική πηγή εγγύηση και διαφάνεια του καταναλωτή. Δηλαδή, η μεγαλύτερη δυνατή σύγκριση μεταξύ ε, προϊόντων επιτρέπει την καλύτερη δυνατή επιλογή. Θα βρούμε λύσεις και για το θέμα του εύρους του ΚΙΤ και το είδος του πληροφοριού που θα περιέχει. Θα πρέπει σε αυτό το επίπεδο να, συνδέσουμε, να συνδυάσουμε από τη την απλότητα με την ανάγκη λεπτομερούς ενημέρωση ώστε να μπορεί να προσανατολίζεται κατάλληλο ο καταναλωτής σε ό,τι αφορά την εναλλακτική επίλυση των διαφορών. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει συνεκτικότητα και ακολουθία με την οδηγία ETR. Πάντως δικό μας καθήκον τη δική μας ε, αυτή η έκθεση είναι να εστιάσουμε στην ευθύνη των κρατών μελών ως εγκύητες της ομαλής διεξαγωγής διαδικασίας και την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή και τη δυνατότητα προσφυγής και μεταξύ αυτών τη δυνατότητα εξοδικαστικής επίλυσης των διαφορών. Τέλος, για την ευθύνη Αντικειμενικά θα έλεγα ότι το παράδειγμα που δόθηκε μεταξύ γιατρού και φαρμακοποιού δεν είναι το πλέον κατάλληλο, γιατί ο γιατρός δίνει μια συνταγή και ο φαρμακοποιός δίνει το φάρμακο, αλλά στην αλυσίδα πληροφόρηση, αν ο ενδιάμεσο έχει και το καθήκον να κατευθύνει προς την αγορά ενός προϊόντος, ε, τότε μια κάποια ευθύνη φέρει ο ε, διάμεσο παραπάνω ευθύνη από ότι ο φαρμακοποιός. Ευχαριστώ πάντως όλους τους ε, συναδέλφους. Πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει πολύ μεγάλη σύγκληση και θα δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Good. Thank you very much all of you for that. Ωραία, σας ευχαριστώ όλους. Και βεβαίω το χρονοδιάγραμμα είναι ανοιχτό προ συζήτηση. Αλλά φαίνεται πω είστε έτοιμο να προχωρήσετε στην ψηφοφορία. Επομένω, ε, η αρμόδια επιτροπή θα είναι αυτή που θα πρέπει να εξετάσει αν θα δεχθεί τι προτάσει μα ε, εγκαίρω ή όχι. Όπως και να έχει. Αυτό είναι δική σας απόφαση. Ωραία. Ευχαριστώ. Ας περάσουμε στο δεύτερο στοιχείο σε αυτό το πακέτο της Επιτροπής ΣΥΤΡΕ. Αναδιατύπωση του Ενωσιακού Τελωνικού Κώδικα. Ο κύριος Κάρας είναι αρμόδιος από το και Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος ε, που τον αντικαθιστά. Α, έρχεται. Στις 11. Ανδιατύπωση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία την άφηξή του. Δεν ξέρω από την άλλη αν είναι εδώ κάποιος. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Η κυρία Ρούλερ, βεβαίως, για τους πρασίνους. Εγώ κατέθεσα κάποιες ε, τροπολογίες από πλευρά CCR. Επομένω, έχει ε, αξιόλογο συνεργάτη εδώ, Κάθριν. Από πλευρά τη Επιτροπή, ε, ποιο είναι μαζί μα, ο κύριο Βανχούλα. Είμαι Στίβεν Ράιαν και αντικαθιστώ τον ε, συνάδελφο. Βεβαίω. Είχα να αλλά δεν ήμουν σίγουρα ποιο ήταν εδώ. Κάθριν Στάιλερ, παρακαλώ. Uh, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και χαίρομαι που έχουμε εκπρόσωπο και τη Επιτροπή. Η πρώτη συνεδρία των Σκιωδών έλαβε χώρα χθε το βράδυ. Θα ήθελα να ευχαριστώ του συναδέλφου για το ενδιαφέρον και για τι προτάσει για τροπολογίε. 182 προτάσει τροπολογιών εν όλο. Ήταν χρήσιμη η χθεσινή συνεδρίαση. Φαίνεται να διαγράφεται συμφωνία σε ορισμένα θέματα, αλλά όχι σε όλα. Στη διαφάνεια, στις ε, διασταυρούμενες πωλήσει δεν φαίνεται να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία, αλλά νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο συνεννόησης προς το συμφέρον των καταναλωτών. Αλλά εάν μπορούμε να συμφωνήσουμε εμείς και αν θέσουμε υπέρ όλων των συμφέρων του καταναλωτού, μπορούμε και σαφές μήνυμα στην Επιτροπή των Οικονομικών Υποθέσεων να αποστείλουμε και ως εκ τούτου να επηρεάσουμε την έκθεση προς την κατεύθυνση αυτή. Η Επιτροπή Έκον την έκθεσή της ουσιαστικά επανέρχεται στο προηγούμενο σύστημα IMD. Ενώ νομίζουμε ότι θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερο, περισσότερη ισχύ, στην, περισσότερη έμφαση στην προσέγγιση του καταναλωτή και να αρχίσουμε από την αρχή το έργο αυτό. Έτσι λοιπόν, και για να απαντήσω στα όσα ακούστηκαν και νωρίτερα και στα όσα προτείνατε, για τον τρόπο να λαμβάνουμε τις αποφάσεις αλλά και να δίνουμε αρκετό χρόνο στην μελέτη των συμβαστικών λύσεων ώστε να έχουμε μια ε, ενωτική λύση και προσέγγιση. Είχαμε αρχικά προβλέψει 20 Μαρτίου την ε, συζήτηση και μέσω μετά την ψηφοφορία. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να καθυστερήσει λίγο η ψηφοφορία, αλλά όπως είπε ο Πρόεδρος, πάλι να έχουμε ένα αποτέλεσμα σαφές ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μπορέσει να επηρεάσει και τις θέσεις της ε- ΕΚΟΝ που αναμένονται για τις 27 Μαΐου. Όσο το δυνατόν πιο ισχυρή λοιπόν τοποθέτηση από πλευρά μα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να δημιουργηθούν πρακτικά προβλήματα αν αλλάξουμε το χρονοδιάγραμμα, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μια μικρή αλλαγή. Και θέλω να ευχαριστώ την Αγγέλικα από την ε, γραμματεία που με βοήθησε και μου έδωσε κατευθύνσει ε, για τι προτάσει μου για την αλλαγή του χρόνου διαγραμματό. Γιατί τελικά νομίζω ότι χάρη σε αυτέ μπορούμε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Όπω είπα, στην απαρίθμιστη διαφάνεια, στην διασταυρούμενε πωλήσει πρέπει να γίνουν ε, κάποιε προσπάθειε παραπάνω για να βρούμε λύσει. Αλλά πάντω από τη χτεσινή μα πρώτη συνάντηση με του Κιώδη, θεωρώ ότι έχουμε περιθώριο να συμφωνήσουμε με λίγο περισσότερο χρονικό περιθώριο θα βρούμε συμβιβασμούς. Και αν τελικά θα τα καταφέρουμε, προτιμώ να έχω στη θέση μου αυτό το επιπλέον διάστημα για να καταλήξουμε σε λύσεις προς το συμφέρον του καταναλωτή, γιατί αυτό που έχει επιλέξει η Επιτροπή των Οικονομικών Υποθέσεων δεν είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τους συναδέλφους για την πολύ καλή συζήτηση χθες. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι για το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να κοιτάξουμε και όλας ε, τι άλλου είδους δεσμεύσεις μπορεί να έχουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, όπως είπατε κι εσείς, το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουν να συναντηθούν, να συζητήσουν και να συμφωνήσουν σε συμβαστικές λύσεις σκιώδεις ηγητές. Είπατε κι εσείς ε, και ο κύριος Παντσέρη έχει καταθέσει ήδη συμβαστικές τροπολογίε, Πιστεύω και εσεί θα τα καταφέρετε. Ναι, Πρόεδρε, η Επιτροπή των Οικονομικών νομίζω ακόμα δεν έχει κάνει καν συνεδρίαση των σκιωδών ε, με τον ε, αρμόδιο κατ' ουσίαν ε, εισηγητή. Ως εκ τούτου εμείς τους έχουμε κάπως προλάβει, είμαστε πιο μπροστά από αυτούς. Καλώς λέω πρόεδρος, θα πρέπει και αυτό να το συζητήσουμε στην προσεχή συνεδρίαση. Ευχαριστούμε, θα δούμε όλες τις προτάσεις και αναλόγως θα διαμορφώσουμε και το χρονοδιάγραμμα για τις λοιπές δεσμεύσεις. Πάντως από τις δύο σας τοποθετήσεις θεωρώ ότι με λίγο περισσότερο χρόνο μπορούμε να ε, εδραιώσουμε τη θέση μα στην τη Επιτροπή των Οικονομικών. Αφού δεν είναι εδώ ο κύριο Καρά, όμω, μήπω να ακούσουμε κάποιον άλλον σκιώδη Γιατί ο κύριο Χατζημαρκάκη, λοιπόν. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Και όντω, όπω και η κυρία Στάιλερ είπε, πολύ σημαντική είναι η ε, συνεργασία που ήδη ξεκίνησε πολύ καλά, πολύ φιλικά και την ευχαριστώ θερμά. Ο στόχος της οδηγίας είναι η διαφάνεια στα ασφαλιστικά προϊόντα υπ' αυτή την έννοια ευπρόσδεκτο. Με τον συνάδελφο Όλυ Σμιτ έχουμε καταθέσει κάποιε προτάσει τροπολογιών και καλώ του συναδέλφου να, την συνάδελφο καλύτερα, να μην λησμονήσει τελείω κατά τη διατύπωση των συμβαστικών τροπολογιών αυτέ μα τι προτάσει. Επί παραδείγματι, στο άρθρο 2 μια τροπολογία μα, όπου ζητούμε ισότιμε συνθήκε ανταγωνισμού, ευκαιρίες ανταγωνισμού για κάθε πράκτορα ώστε να έχει και την ίδια προστασία του καταναλωτή. σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να επιδιώκει η οδηγία. Το έχουμε καταγράψει τροπολογία. Επίσης, για την ελευθερία της εγκατάστασης έχουμε καταθέσει δύο τροπολογίες και την ελεύθερη κυκλοφορία του πράκτορα των ασφαλίσεων, του διαμεσολαβητή αν θέλετε. Είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία. και τα άρθρα 3 και 6 συγκεκριμένα οι τροπολογίες, εκεί που αναφέρεται η ελευθερία της εγκατάσταση. Έχουμε επίση τροπολογία ως προς την ε, παροχή συμβουλών, που γνωρίζουμε και από τις τράπεζες. Όταν ε, πάει κανείς να αισθήσει ε, δάνειο γίνεται μια συζήτηση. Το έχουμε ζήσει όλοι πιστεύω αυτό με τον εκπρόσωπο της τράπεζας. Αλλά βέβαια ξέρουμε ότι ανάλογα με το κράτος μέλος έχουν διαφορετικές πρακτικές. Φερρυπίν, εάν ε, είναι υποχρεωτική υπογραφή του υποψηφίου πελάτη ε, ότι έλαβε την ενημέρωση και την κατάλαβε σωστά. Μπορεί να διαφέρει σαν υποχρέωση από, την άλλη, από τη μία χώρα στην άλλη. Ε, αντίστοιχα λοιπόν ένας κατάλογος των στοιχείων που θα πρέπει να διατίθενται, των πληροφοριών δηλαδή, που θα πρέπει να μπορεί και ο πελάτης να παρακολουθήσει, να αντιληφθεί και βέβαια η συζήτηση αυτή θα πρέπει να γίνεται με τον κάθε πελάτη και εμείς λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα τυποποιημένο κατάστοιχο, ένας κατάλογος τυποποιημένος των πληροφοριών των σχετικών με την ασφαλιστική σύμβαση που θα πρέπει να λαμβάνει στην πραγματικότητα ο υποψήφιος πελάτης. Και το άλλο ζήτημα είναι αυτό της ελάχιστης εναρμόνισης. γιατί με κάθε σεβασμό βέβαια προς την ε, ομοιομορφή ρύθμιση δεν μπορούμε και να ε, αφαιρέσουμε κάθε τύπου ελευθερία στα κράτη-μέλη και γι' αυτό στην, ε, στο άρθρο 19 καταθέτουμε μια πρόταση τροπολογία για ελάχιστη εναρμόνιση. Σε ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ράιαν που θα ήθελε να σχολιάσει αυτά τα ζητήματα και βεβαίω όταν έρθει ο κύριο Κάρα θα του δώσω το λόγο. Αλλιώ μπορούμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μερικέ ε, γενικέ παρατηρήσει και μετά ορισμένα πιο συγκεκριμένα ζητήματα για τι προτεραιότητε τη Επιτροπή. Πρώτα απ' όλα, σαφώ και πρόκειται για μια πρόταση που ε, προσανατολίζεται προς τον καταναλωτή και μπορούμε να την εξετάσουμε μόνο στο ε, πλαίσιο των πακέτων όπως το PRIPS που συζητήσαμε πριν λίγο και το MIFID. Ο παραλληλισμό με το MIFID είναι εξαιρετικά σημαντικό, εφόσον ε, ε, ε, το πακέτο MIFID συμπεριλαμβάνει και του κανόνε πώληση των μη ασφαλιστικών πρίψ και αυτή εδώ η πρόταση συμπεριλαμβάνει τα, και τα ασφαλιστικά πρίψ. Οποιαδήποτε απόκληση μεταξύ των δύο στο τέλο τη διαδικασία διαμεσολάβηση μπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό ο παραλληλισμό. Ε, συμπληρώνουν, συμπληρώνονται κάποια από τα κενά του πρώτου ε, IMD σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή. Ε, αυξάνει το επίπεδο προστασία των καταναλωτών, ενώ παραμένει ελάχιστη αναρμόνιση. Οποιοςδήποτε έχει εξετάσει την εξολόγηση δικτύπου θα δει ότι ε, σαφώς πήραμε υπόψη το ζήτημα του άχθους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νομίζω ότι έχουμε βρει την κατάλληλη ισορροπία σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών και το άχθος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, για κάποια πιο συγκεκριμένα σημεία. Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής εδώ. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή, θέλουμε να παραμείνει ευρύ αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και κάποιες ε, κάποιους τομείς όπου υπάρχουν ε, καταχρήσεις. Ε, αυτό συμπεριλαμβάνει τα ταξιδιωτικά γραφεία, όπου υπήρξαν παραπλανητικές πωλήσει και άλλοι τομείς. Και δεν θα θέλαμε να ε, εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογή τέτοιου είδους τομείς. Γιατί ακριβώς για αυτές τις για αυτούς του τομεί υπάρχει αυτή η πρόταση. Άλλος ε, κύριος στόχο είναι η διευκόλυνση των διασυνοριακών πτυχών ε, τέτοιων υπηρεσιών. Όμω αυτό θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή τη αμοιβέ αναγνώριση, που βασίζεται και σε πολύ εύρωστο ορισμό των ελάχιστων ε, επαγγελματικών προσόντων που απαιτούνται. Μπορούμε να συζητήσουμε ποια είναι αυτά τα ελάχιστα επαγγελματικά προσόντα, όμω είναι κύριο ε, στοιχείο της διασυνοριακής αμοιβές αναγνώρισης ε, και οι προϋποθέσεις συνεχιζόμενης κατάρτισης. Θεωρούμε ότι ένα, μια κατάλληλη μέθοδος για τον προσδιορισμό των λεπτομεριών θα είναι η καταξιδότηση πράξης της Επιτροπής. Προφανώς δεν συμφωνούν όλοι με αυτό, το κατανοούμε. Όμως οι λεπτομέρειες είναι σημαντικές. Για παράδειγμα για τα επαγγελματικά προσόντα. Και αν αποφασίσουμε να τα εντάξουμε στην βασική οδηγία, τότε θα πρέπει να υπάρχουν ε, μακροσκελείς ε, συζητήσεις με τους πραγματογνώμονες, ενώ θεωρούμε ότι η κατεξουσία της πράξης είναι ένα πιο κατάλληλο μέσο. Και τέλος, ο παραλληλισμός ε, με την οδηγία για το εργαλείο αγοράς ε, θα είναι κάτι που θα μας ε, βοηθήσει ιδιαίτερα με άλλα στοιχεία για τη διασταυρούμενη πόλη, για παράδειγμα. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να αντιλήσουμε έμπνευση από αυτή την οδηγία τη ΜΥΦΙΤ για τέτοια στοιχεία. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες εδώ. Όμως ελπίζω αυτές ε, οι παρατηρήσεις κάπως να λειτουργήσουν διευκρινιστικά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, περιμένουμε ακόμα τον κύριο Κάρας. Είναι εδώ ή όχι. δεν μπορούμε να ε, σχεδιάσουμε συνεδριάσεις γύρω από τη διαθεσιμότητα των σκιωδών. Οπότε θα δώσω το λόγο και πάλι στην εισηγήτρια να κλείσει. Ίσως αν το πάτε ως 11, να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Κάρας να σα ξαναδώσω πάλι το λόγο, εισηγήτρια. Αρκεί και να δώσω το λόγο στον κύριο Φόξ ακριβώς. Δεν ξέρω, πρόεδρε, μου χρειάζονται πέντε λεπτά. Ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που ακούσαμε από την Κομισιόν. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική αυτή η πρόταση, ιδίω λόγω των παρελθόντων στοιχεία με το MIFID. Γι' αυτό και εμείς το επισημάναμε. Παράδειγμα, όταν η Επιτροπή μιλά για τη σημασία να συμπεριλάβει τα ταξιδιωτικά γραφεία. Η ΕΚΟΝ το διέγραψε. Διέγραψε τους ε, ταξιδιωτικούς πράκτορες από την πρότασή της. Ε, αυτό υπονομεύει σημαντικά τον αρχικό στόχο οι διαφωνίες λοιπόν που υπάρχουν πολλέ φορές σε άλλα θέματα όπως οι υπεσχρωσιοδότες είναι αστείες σχέση με αυτά τα θέματα όπως είναι οι διαστηριακέ ε, υπηρεσίες κτλ. Έτσι εν κατακλείδη θα έλεγα ότι αν είχαμε ελαφρά ένα μεγαλύτερο χρονοδιάγραμμα ώστε να μπορέσουμε να ξαναδούμε κάποιες συμβατικές τροπολογίες λαμβάνοντας πάντοτε ως γνώμονα τον καταναλωτή. Γιατί και πάλι αν δεν κάνω λάθος 22 Μαΐου ψηφίζει η Επιτροπή ΕΚΟΝ. Αν λοιπόν πριν έχουμε ενοποιημένη θέση, τότε θα ενισχυθεί η θέση μας και θα δείξει τη σαφή διαφορά στην προσέγγιση ανάμεσα στις δύο επιτροπέ. Το χρονοδιάγραμμα βεβαίως εξαρτάται από τους συντονιστέ και από ό,τι μας δώσετε τελικά. Πάντως ευχαριστώ τους σκιώδεις και ελπίζω να καταλέξουμε σε έναν ισχυρό συμβιβασμό και στον τομέα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα ξαναδούμε το χρονοδιάγραμμα και για τις δύο προτάσεις και θα είναι αρκετά πυκνό το πρόγραμμά μας στο επόμενο διάστημα και δεν μπορώ να σας το εγγυηθώ. Γιατί θα εξαρτηθεί και από την ψηφοφορία και από τι βασικέ τροπολογίε, οπότε είναι κάπω ένα φαύλος κύκλο. Ευχαριστώ όλου. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Ένα σύντομο διάλειμμα για καφέ. Παρακαλώ όμως να είστε ακριβώ εδώ στι 11 και 10 για να ξεκινήσουμε αμέσω την πρόταση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε νωρίτερα γιατί θέλω να είναι άπαντες παρόντες. Παρακαλώ να είσαστε εδώ ακριβώς την ώρα σας. Και Κάρας, λυπάμαι, αλλά οι πολιτικές ομάδες και όδης εισηγητές σε κάποιο λόγο. Για να είναι και παρόντες θεδριάσεις. Το χρονοδιάγραμμα, μάλλον το πρόγραμμά μας ήταν στη δίθεσή σας πολύ νωρίτερα. Δεν γίνεται δεν γίνεται αλλιώς και δεν είναι καθόλου ωραία εικόνα στο κοινό ε, να μην εκπροσωπούνται συζητήσεις τα, οι μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες. Θεωρώ ότι αυτό είναι ευθύνη των πολιτικών ομάδων. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη αν ήμουν έτσι κάπως αυστηρός το, το πρωί. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε ακριβώς στις 11 και 10. Uh, Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που επιστρέψατε στην αίθουσα εγκαίρως. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για, την, τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και να καλωσορίσω ιδίω όσου μας παρακολουθούν μέσω web streaming για αυτό ακριβώ το σημείο. Να υπενθυμίσω και στους που βλέπετε το διαδίκτυο αυτό το newsletter που μπορείτε να λάβετε κι εσείς αν το ζητήσετε μέσω email. Θα δείτε στο website μας το email, όπου εκεί μπορείτε να μας αποστείλετε το εκτιμά σας και κάθε μήνα θα λαμβάνετε αυτό το εφημεριδάκι. Λοιπόν, με μεγάλη χαρά να ξεκινήσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση για την έκθεση πρωτοβουλίας της Επιτροπής μας, ανταποκρινόμενη στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Είναι ένα θέμα μας απασχολεί εδώ και χρόνια στην Επιτροπή μας. Υπάρχει πλέον μια κάποια εμπειρογνωμοσύνη και θα και η κυρία Πατίνη είναι να γνωρίζουν ιδιαίτερα το θέμα. Δεν συμφωνούμε πάντοτε, αλλά πιστεύω ότι η γνώση θα οδηγήσει βαθμία στην συμφωνία. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου. Ο κύριος Ασχληφόξ θα πάρει το λόγο θα τον καλέσω να μας παρουσιάσει εντάχει τις προτάσεις του, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πάρουν το λόγο, όλοι οι συναδελφοί, εδώ, όλοι όσοι έχουν εμπειρία του θέματος, πέρα από τους κοιόδης για αυτό το θέμα, ο Χαριτίνινγκ επίσης ως αναπληρωτής επικεφαλής μονάδας και ο Χόγκαν επίσης Justice Officer για αυτό το φάκελο. Οπότε, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, δίνω το λόγο στον κύριο Φόξ. Πάντως θα πρέπει να κλείσουμε ακριβώς πριν τις 12. Έχουμε τρία τέταρτη θέση μας, οπότε σε αυτή τη φάση μπορούμε να είμαστε λακωνικοί, γιατί θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες στο μέλλον. Κύριε Φόξ, παρακαλώ, μπορείτε να ξεκινήσετε τη ζήτηση για αυτή τόσο σημαντική ε, έκθεση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για το διορισμό μου ως εισηγητή σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Είναι σημαντικό όχι μόνο για τη δική μου ε, περιοχή από που προέρχομαι, αλλά και την ενιαία αγορά. Και χαίρομαι γιατί γιατί συνεργάζομαι με δύο πρώην εισηγητέ που έχουν οριστεί τώρα και η γνώση του, ε, μαζί με όλους όλους σκιώδες είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα. Είδαμε ότι αυτή η Επιτροπή να προχωρά από την έκθεση Σάτμακερ και Κρόιτσερ και πάμε τώρα στη δική μου. Και ελπίζω με... να διατηρήσουμε το κολέκτηρο συνεργασία μεταξύ των ομάδων. Τι τελευταίε εβδομάδε έκανα μια συντονισμένη προσπάθεια να συναντήσω όλου του ενδιαφερόμενου φορεί φορείς, εμπορικούς, αριθμιστικές αρχές, αθλητικούς φορείς, ρυθμιστικούς φορείς και άλλες ε, ομάδες ε, άσκησης πίεσης και ενδιαφέροντος. Το θέμα του διδεκτικού ε, τυχερών παιχνιδιών είναι κάτι διασυνεριακό και είναι σε ένα βαθμό κάτι που μπορούμε να δώσουμε μια εναρμόνιση στην εσωτερική αγορά. Βλέπετε όμως τι συμβαίνει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, τηρώντα και την αρχή της επικουρικότητας, βεβαίως, στο βαθμό του δυνατού. Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να σα παρουσιάσω τους γενικούς τομεί που θα θίξω στην έκθεσή μου, ξεκινώντα ε, απευθύνοντας ευχαριστίες προς την Επιτροπή, γιατί έχει υποβάλει μια καλή ε, πρόταση που είναι μια καλή βάση για εργασία. Ο πρώτος τομέας που πρέπει να αναλάβουμε δράση είναι η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οι πιο πολλοί συνάδελφοι θεωρούν ότι πλέον έχει περάσει αρκετός καιρός όπου ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κάνει ελάχιστη ως τίποτα για να εφαρμόσει το ε, κοινοτικό δίκαιο. Κάτι πολύ θλιβερό και ιδίω με τη δημοσίευση της έκθεσης Κρόιτσμαν η Επιτροπή έχει αναλάβει μια πιο ενεργητική, αν θέλετε, στάση. Μπορεί να κάνει όμως πιο πολλά ακόμη και την καλό να εφαρμόσει τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Η ενιαία αγορά, εσωτερική αγορά, θα αποφεληθεί από τη διοικητική συνεργασία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών για θέματα επιβολής. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε κοινά τεχνικά πρότυπα ώστε να μεσούμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Τι εννοώ για παράδειγμα. Ένα κοινό, μια κοινή ταυτοποίηση των παικτών ένα πρακτικό τομέα όπου μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια προστιθέμενη αξία. Έπειτα, πρέπει να λάβουμε δράση στο τομέα προστασία καταναλωτή και στον τομέα τη διαφήμιση. Παράδειγμα, να μπορεί ο καταναλωτή να θέτει όρια στα παιχνίδια ή να αυτοαποκλείεται από συγκεκριμένα site και αυτό να μπορεί να ισχύει για όλη την εσωτερική αγορά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με ένα α, κώδικα να θέσουμε κάποια όρια που θα πρέπει να ε, υποχωρεούνται οι πάροχοι να παρουσιάζουν στην οθόνη και ε, ανάλογα, αν δεν υπακούν και με τον κώδικα διοντολογίας, να ε, υπάρχουν και πιο αυστηρές κυρώσεις. Ή Επίσης να διασφαλίσουμε και την ακαιρεότητα του αθλητισμού, ώστε τα διδακτικά τυχερά παιχνίδια δεν είναι δεν εμπλέκεται σε στιμένους αγώνες και άλλες κλιματικές πράξεις. Η έκθεσή μου θα είναι έτοιμη ως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Οι σκιώδες θα λάβουν να γραφώ στα αγγλικά και με, αμέσως θα περάσει και σε μετάφραση ε, η πρότασή μου. Θέλω να ακούσω τώρα από τους άλλους σκιώδεις τις απόψεις τους. Ε, θέματα, ευρύτερα θέματα, θεματικές ενότητες που έχω α, παραλείψει και παρακαλώ πείτε, τα τα μου για να τα συμπεριλάβω στο πρώτο σχέδιο. 4 Απριλίου υποβολή τροπολογιών και ελπίζω ότι ως τότε να έχω τη συνάντηση με τους κοιόδες για να συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την ευρύτερη δυνατή συνένεση. Κλείνοντας λοιπόν, λέω ότι προσβλέπω σε καλή συνεργασία πρόεδρε μαζί και με τους άλλους κοιόδες για να καταλήξουμε σε μια έκθεση που λαμβάνει υπόψη όλες τις απόψεις αυτής της Επιτροπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ξεκάθαρη παρουσίαση των βασικών σημείων της εκθέσης. σας, κυρία Πιτικά είναι να θα ξεκινήσει τη συζήτηση εξ ονόματος των σκιωδών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την πολύ επικοδηματική του εισαγωγή και την προθυμία του να συνεργαστούμε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι αναγνωρίζω απολύτως ότι πρόκειται για ένα λεπτό ζήτημα. Τα κράτη-μέλη έχουν επιλέξει διαφορετικές ε, προσεγγίσεις από ιδιαίτερα φιλελεύθερες έως ε, πολύ περιοριστικές έως και μονοπωλιακές. Αυτή την αρχή πρέπει να την ε, αποδεχθούμε και να τη σεβαστούμε και πρέπει να την ε, δεχθούμε ως μία φωτηρίας. Προσωπικά και εκ μέρους της ομάδας μου σας διαβεβαιώ ότι θα προσπαθήσω να εργαστώ στο δυνατόν με περισσότερο διαφανή ξεκάθαρο και ανοιχτό τρόπο για να συγκεράσουμε διαφορετικές γνώμες, γιατί θεωρώ ότι αυτό θα αποβεί σε όφελος των καταναλωτών. Αν δηλαδή υπάρξει μια κοινή άποψη και γνώμη για αυτά τα ζητήματα, συμφωνώ ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι μάλλον εξισορροπημένη και το ζήτημα αυτό των τυχερών ε, παιχνιδιών στο διαδίκτυο ε, είναι εγγενώς ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο ζήτημα. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ε, εξισορροπούμε τα εξή δύο ζητήματα. Αφενός τη δραστηριότητα που είναι εγγενώς ευρωπαϊκή και παγκόσμια και έτσι απαιτεί αντίστοιχες δράσεις και αφετέρου τις πολύ διαφορετικές στρατηγικέ και πολιτικέ που ακολουθούν τα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να σεβαστούμε. Πρώτη μου παρατήρηση είναι ότι ο τζόγο τα τυχερά παιχνίδια έχουν ε, έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Δεν μπορούν να συγκριθούν με άλλα προϊόντα στην εσωτερική αγορά των υπηρεσιών. Μπορεί να συγκριθεί ε, με άλλα προϊόντα απόλαυση των εισαγωγικών όπως το αλκοόλ και, τα... και ο καπνός και εκεί μπορούμε να, θα μπορούσε να υπάρξει απαγόρευση και να συμβαίνει όλο το εμπόριο αυτό παράνομα και αυτό να δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα. Όμως, ε, χάρη εξαιτίας μάλλον της εθιστικής του φύσης, πρέπει να ρυθμίζεται πολύ στενά και να αναγνωρίζεται ο ειδικό του χαρακτήρα. Μετά έχουμε το υψηλό επίπεδο προστασία καταναλωτών, ε, προστασία των ανηλίκων, προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που πρέπει να είναι ο δεύτερο μεγάλο στόχο μα. Πού μα οδηγεί αυτό, Έχουμε προβλήματα που συνδέονται με το ξέπλυμα πνευματικού χρήματο, με τι εγκληματικέ δραστηριότητε, ε, εθισμού και άλλες προβληματικές καταστάσεις. Και αυτές οι καταστάσεις φαίνεται ότι επικεντρώνονται περισσότερο στις διαδικτυακές ε, δραστηριότητες παρά στις φυσικές. Τι κάνουμε λοιπόν και πώς προστατεύουμε τον παίχτη. Πρώτον, χρειάζομαστε ε, μία ένα νομικά δεσμευτικό σύστημα ταυτοποίησης ε, με στεγανά για τον παίχτη. Πρέπει να δημορφώσουμε ένα σύστημα όπου υπάρχει ταυτοποίηση του παίχτη και περιορισμένος αριθμός ε, είτε αριθμών πιστοτικής κάρτας, είτε τραπεζικών λογαριασμών, οτιδήποτε και αν συμβαίνει, για να εντοπίζουμε τον παίχτη από πού έρχονται τα χρήματα και πού πηγαίνουν. Και βλέπετε ότι αυτό συνδέεται και με το ξέπλυμα χρήματο, με άλλε εγκληματικέ δραστηριότητε, με την απόδοση φόρων ε, στην ε, συναφή χώρα και το καθεξής. Δεύτερον, μετά αυτή την ταυτοποίηση θα πρέπει να υπάρχει ένα ε, ένα, όριο που θέτει ο, ίδιος ο παίχτης στον εαυτό του και ένας αυτοαποκλεισμός ε, ε Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά είναι εφικτό. Ουσιαστικά θα πρέπει όμως να έχουμε ένα κοινό σύστημα ή δεξαμενή, όπου ο, ε, ο παίκτης μπορεί και θα πρέπει, θα, θα πρέπει να είναι αποχρεωμένος να, αποδεχθεί ότι όταν ε, ξεπεράσει το όριο παιχνιδιού και μετά μπλοκάρετε. Όμω βέβαια αυτό δεν έχει νόημα. Αν μπορεί κάποιο να φτάνει μεν στο όριο σε ενα, ιστότοπο, αλλά μπορεί να πάει σε ένα άλλο μέχρι να φτάσει και εκεί το ε, όριο. Επομένω θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών και να τηρούνται τα όρια. Και τα δύο αυτά ζητήματα θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τα τευθυντήριες γραμμές. Τρίτο σημαντικό στοιχείο. Μακροπρόθεσμα, για να γίνουν αυτές οι ενέργειες πραγματικά νομικά δεσμευτικές και για τους παρόχους υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά, θα πρέπει η παραγωγή, οι πάροχη των υπηρεσιών να καταχωρίζονται στην Ευρώπη ή να έχουν λάβει κάποια διοδότηση; Δεν μπορούμε να έχουμε όλους τους εθνικούς μηχανισμούς ακυρώσεων και να είναι δεσμευτικοί αν δεν υπάρχουν σε κάποιο μητρό, αν δεν έχουν καταχωριστεί. Τέλος, για την μη δίκαια διαφήμιση και μετά υπάρχει το ζήτημα της ε, συμμόρφωσης με το ρυθμιστικό, του ρυθμιστικού πλαισίου με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Όπως είπε και ο συγητής, πρέπει να ενταθεί και να ενισχυθεί η διοικητική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ωραία. Σα ευχαριστώ πολύ για τι σαφέ σας προτάσεις, κύριε Σαντερμόσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Φόξ, για την παρουσίασή σας. Είναι ενδιαφέρον ζήτημα, το συζητούμε και πάλι. Είναι σαφές ότι προοδεύουμε στις συζητήσεις μας και αυτό είναι απαραίτητο. Εκ μέρου ε, των ε, Σοσιαλδημοκρατών, ε, πραγματικά χαιρετίζουμε την ανακοίνωση τη Επιτροπή, την επικροτούμε. Είναι μια καλή ανακοίνωση. σχολιάζει και του απαραίτητου τομεί, όπως είναι οι στημένοι αγώνες. Είναι σημαντικό πρόβλημα και θα πρέπει κάτι να κάνουμε σε αυτό. Αυτό που λείπει όμως από την ανακοίνωση είναι η Επιτροπή επιτέλους αναγνωρίζει ότι χρειαζόμαστε μια σταδιακή ε, διαδικασία. Δεν μπορούμε να κινηθούμε πολύ γρήγορα. Πρέπει να αποδεχθούμε τις ε, ε, πολιτιστικές ή πολιτικές διαφορές των κρατών μελών, να σεβαστούμε την αρχή της επικουρικότητας. Πέρα από αυτό όμως, θεωρώ ότι μπορούμε να προοδεύσουμε σε ό,τι αφορά την προστασία καταναλωτών. Γιατί προφανώς και θέλουμε και πρέπει να προστατεύσουμε τους καταναλωτές, ε, τους παίχτες και τα ανήλικα. Και δεν θεωρούμε ότι το κάνουμε αυτό σε ικανοποιητικό βαθμό. Θα το εξετάσουμε λοιπόν κατά τη διάρκεια της ε, εξέτασης πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα επίπεδα προστασία των καταναλωτών. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανησυχία των σοσιαλιστών. Όμως δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω ότι χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό για, το, για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια. Όμως ό,τι αφορά τη διοικητική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών, ε, πράγματι μπορούμε να προοδεύσουμε. Ε, συμφωνώ με την ε, ομάδα εμπειρογνωμόνων που ξεκίνησε την Επιτροπή. Ίσως μπορούμε να βρούμε και κάποιες ιδέες για το πώς μπορεί να βελτιωθούν οι εργασίες της. Όμως θεωρώ ότι πρέπει να συζητήσουμε και βεβαίως να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Πρέπει όμως να πω ότι είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανείς με τον κύριο Φόξ όταν λέει ότι πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς νόμους. Ε, δεν μπορεί βεβαίως κανένας να ε, φέρει αντίρρηση. Όμως, παράλληλα, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι πρέπει να γνωρίσουμε ότι τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο δεν είναι μια φυσιολογική συνήθιση οικονομική δραστηριότητα. Έχει, έναν, έχει ειδικά χαρακτηριστικά. Και έτσι ο τομέα πρέπει να συμμορφούνται με όλη την νομοθεσία και του κανονισμού για την εσωτερική αγορά. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα ειδικά χαρακτηριστικά. Όπω ε, συμβαίνει και με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρέπει λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία. Αναγνωρίζουμε βεβαίω ότι έχει ειδικά χαρακτηριστικά αυτό ο τομέα των τυχερών παιχνίων και μετά να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε αυτό το, αυτή την προϋπόθεση, ότι πρέπει δηλαδή να συμμορφούνται και με τις αποφάσεις του δικαστηρίου και με την ομοθέσια εν γέννη. Κάτι που θεωρώ θετικό και συνέβη στα κράτη-μέλη το τελευταίο διάστημα είναι ότι υπάρχουν εξελίξεις, ε, κράτη-μέλη ανοίγουν τις αγορές τους και πρέπει να αποδεχθούμε ότι θα μας πάρει ένα χρονικό διάστημα αυτή η διαδικασία και πρέπει να βρούμε τον τρόπο που ταιριάζει και στο κάθε κράτο μέλος. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση λοιπόν είναι η πλέον κατάλληλη. Στη Δανία, επί παραδείγματι, έχουμε μια νέα αρκετά φιλελεύθερη ε, νομοθεσία για τα τυχερά παιχνίδια και Όταν ε, συνομιλώ με εκπροσώπους του χώρου εδώ, πολλές φορές ε, μου λένε τι θετική εμπειρία έχουν ε, από το δανεικό παράδειγμα, γιατί είναι πολύ ανοιχτό το σύστημα, είναι εύκολο κανείς να πάρει μια άδεια. Όμως, κατά τη γνώμη μου, δεν λειτουργεί καλά το σύστημα. Είναι πράγματι εύκολο να πάρει κανείς άδεια, όμως δεν μπορεί να ανοίξει κανεί μια εφημερίδα, έναν ιστότοπο ή να παρακολουθήσει μια ταινία στην τηλεόραση χωρίς, χωρίς να πέσει πάνω σε μια διαφήμιση για τα τυχερά παιχνίδια. Και αυτό είναι εξαιρετικά επιθετική πολιτική, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό θα πρέπει, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Να έχουμε μια ανοιχτή αγορά βάσει για τον αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, αλλά τότε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το γεγονός ότι δεν μπορούμε να έχουμε τους ίδιους κανόνες ε, διαφήμισης ε, όπως με όλους τους υπόλοιπους τομείς. Ε, τα παιδιά μου, ας αγαπούν το ποδόσφαιρο. Βλέπουν την Bayern, για παράδειγμα, ναι, πράγματι, αλλά ε, κάθε φορά που βλέπουν έναν αγώνα, πέφτουν πάνω σε διαφημίσεις για πόκερ και άλλα παιχνίδια. Για μένα είναι πρόβλημα αυτό και πρέπει πραγματικά κάτι να κάνουμε κάτι για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Σε αυτό το σημείο λοιπόν είμαι ανοιχτή προς συζήτηση. Υπάρχουν πολλά όμως σημεία πρέπει να συζητήσουμε, θα μείνω εδώ. Προσβλέπω όμως ε, ε, στη συνεργασία μας και στις συζητήσεις μας τις επόμενες εβδομάδες και σίγουρα θα καταλήξουμε σε μια καλή λύση στο τέλος. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Είναι ήδη ξεκάθαρο, κάτι που σημαίνει και στην αρχή, ότι ήδη έχουμε βαθιά γνώση από πλευρά κάποιων συναδέλφων σε αυτό το τομέα. Είναι καλό λοιπόν να βασιστούμε σε αυτή τη γνώση. Και ξέχασα να φέρω κάποιου πριν, όπω ο κύριο Κρότσμαν, που εκπώνησε τη δεύτερη ε, έκθεση μετά τη κυρία ε, Σαντλεμότσε. Παρακολουθώ και το λόγο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα κάνω ένα σχόλιο στα αγγλικά όλοι λέμε κάτι για την αρχή της επικουρικότητας. Ναι, συμφωνώ, αλλά η λύση δεν μπορεί να έρθει μόνο από την Ευρώπη για να προστατεύσουμε ευάλωτα πρόσωπα, τον εθισμό, ε, το στήσιμο παιχνιδιών, το ξέπλυμα ευρωπαϊκού χρήματο. Αυτό δεν λύνεται σε εθνικό επίπεδο. Και είναι ξεκάθαρο. Φυσικά η διαδικασία θα είναι βαθμία, δεν υπάρχουν συστήματα διοδότησης σε όλες τις χώρες. Η Δανία είναι χρηστική και ενδιαφέρουσα περίπτωση. Και το γερμανικό μοντέλο το ξέρετε γιατί περιορίζεται σε 20 μόνο παρόχους. Αλλά είτε το πείτε ρυθμισ... ρυθμίσεις, ρυθμιστικό πλαίσιο, είτε το πείτε με κάποιο άλλο όνομα, ε, πρέπει να βρούμε μία λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λέει ότι όσο πιο πολλέ άδειε έχει μια εταιρεία, τόσο μεγαλύτερη προστασία του καταναλωτή. Αυτό κατάλαβα από την τελευταία απόφαση του ΔΕΚ. Όταν έχεις και γκρίζα και μαύρη αγορά, πώς θα το τον καταναλωτή. Όταν υπάρχει ένα σύστημα αδειοδότησης, εκεί μπορείς να ορίσεις πρώτα απ' όλα ποιο και πώ μπορεί να πάρει άδεια. Τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα και μετά μπορεί να απαγορεύσει κάποια πράγματα και να επιστρέψω στα γερμανικά. Γιατί το τοποθέτησαμε στα γερμανικά. Με την ε, πρωτοβουλία αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί μια ευρεία έκκληση για συνεργασία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακούσαμε το κυρία <coughs> Ντεμόζο ε, θεωρώ ότι οι περισσότερες προτάσεις εκθέσεως μου καταγράφονται στο, πιστεύω πρόγραμμα δράσης. Πιστεύω πάντως ότι η πρωτοβουλία δεν είναι αρκετά θαραλέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εύστοχα να γνωρίζει ότι χρειάζεται ένα ευρύ πλαίσιο ρυθμιστικό ώστε να προσδιοριστούν τα όρια της εσωτερικής αγοράς, να παρεμποδιστεί η διάπραξη εγκλημάτων και να διαφυλαχθεί και η ακαιρεότητα του αθλητισμού. Σε μια αγορά ψηφιακή χωρί όρια. Αυτό δεν μπορούν να το επιτύχουν μόνο του τα κράτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφει ορθά τα, τα, προβλήματα, δεν προσφέρει όμω επαρκεί λύσει. Και ιδιαίτερα το πρόγραμμα δράση δεν περιλαμβάνει καμία πρόταση για δεσμευτικά νομοθετήματα σχετικά με, το με τη διαδικτυακή χορτοπεξία. Απλώ προσπαθεί με ε, μη δεσμευτικέ συστάσει και ε, παροτρύνσεις να λιδώσει λύσεις σε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Πιστεύω ότι χρειάζονται περαιτέρω ε, νομοθετικές προτάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταλήξει ασφαλώς ε, εν τέλει στο συμπερασμό ότι πρέπει να κάνει ένα βήμα παραπάνω προς την κατεύθυνση αυτή. Ελπίζω να έχει κάθε επιτυχία στην εφαρμογή των αρχών της ιστορικής αγοράς και στα θέματα αυτής της ηλεκτρονικής χαρτοπεσίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάνω απ' όλα να πείσει για τη σημασία του στα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη το Κοινοβούλιο πάντοτε επιμένει στην ε, ανάληψη της υπευθυνότητα και των ευθυνών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής ω στρατοφύλακα των συνθήκων και θα πρέπει να αναλάβει τα δράσει σε περίπτωση που τα κράτη-μέλη δεν προσφέρουν επαρκώς και εγκαίρω ε, πληροφορίες για την εθνική του νομοθεσία, για την συνεργασία μεταξύ των διοικητικών αρχών που προτείνει επίση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ότι στόχο θα είναι να αποφευχθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να διευκολυνθεί η προστασία του καταναλωτή. Ναι, αλλά δεν δίνονται λεπτομέρειε. Δηλαδή, μπορεί για χάρη τη προστασία του καταναλωτή να διατηθέται πληροφορίε για ε, προσωπικά δεδομένα και ε, για την υπόλοιπη λειτουργία της αγοράς. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι μπορεί να γίνει βελτίωση των ε, στοιχείων που θα προσφέρονται. Ε, η προστασία του καταναλωτή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πιστεύουμε ότι απαιτούνται ισορροπημένες ε, συνθήκες πλαισίου για να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, αλλά ε, δεν μπορούν μόνο οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις να οδηγήσουν σε αποτελέσματα όταν δεν υπάρχει επαρκή προστασία του καταναλωτή από τους ε, άπλιστους κερδοσκόπους. Και γι' αυτό νομίζω ότι, θέλουμε, ότι χρειάζονται πολύ πιο ε, ευρείες ρυθμίσεις συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για την αντιμετώπιση της ε, χαρτοπεξίας, εθνικών αστυνομικών αρχών και των διεθνών διοκτικών αρχών, πράγμα το οποίο θα σήμαινε για ορισμένα κράτη-μέλη ή γενικότερα για τα κράτη-μέλη και την θέσπιση θέσεων συνδέσμων ή σημείων επαφής ή αξιωματούχων επαφής και εδώ θα πρότεινα ε, την παρατήρηση ότι και η απάτη όσο και η νομοποίηση παρανόμων εσόδων θα πρέπει να αναγνωριστούν ως παράγον επιδείνωσης κατάστασης. Θα πρέπει λοιπόν οι προδιαγραφές για την χαρτοπεξία να ξεκαθαριστούν και η πρόταση είναι πολύ καλή. Η πέμπτη προτεραιότητα για τη διαφύλαξη της εκαιρεότητας του αθλητισμού και την ε, αποτροπή των κερδοσκοπικών κινήσεων και της χειραγώγης παιχνιδιών είναι πολύ σοβαρός στόχος και πιστεύω ότι θα πρέπει και οι αθλητικοί σύλλογοι και οι αρχές να συνεργαστούν στενά για να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους αλλά και με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές διώξεως όπως Ευρωπολ και Ιντερπολ ε, ώστε να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα χειραγώγησης παιχνιδιών. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Περιμένω να δω τις προτάσεις του συναδελφού Φόξ και Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία για να εξασφαλίσουμε ευρύτατη βάση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι με την έκθεση αυτή μπορούμε να εξασφαλίσουμε την υποστήριξη τη συντριπτική ε, πλειοψηφία των κρατών βουλευτών μα, ώστε να ενθαρρύνουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πιο αποφασιστική δράση. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ε, επιλύσουμε τα προβλήματα σε ευρωπαϊκή βάση δηλαδή. Και άρα θα πρέπει να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την ενθαρρύνουμε διαφορετικά ώστε να προχωρήσει πολύ πιο φασιστικά με διαφύλαξη φυσικά τη αρχή τη ε, επικουρικότητα, να ρυθμίσουμε τα πάντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε πολύ σοβαρή δουλειά στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Κυρία Ρούλερ και μετά Βουγγέζη. Ευχαριστώ. Δεν ευχαριστώ βέβαια τον εισηγητή γιατί δεν έχουμε πρόταση, αλλά τον κύριο Χρόιτσμαν ιδιαίτερα. Η δική του η έκθεση έχει εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Μπορούμε να στηριχθούμε σε αυτήν για να την αναπτύξουμε και πιστεύω ότι θα ήταν σκόπιμο ο κύριο Φόξ να στηριχθεί στη δική σα έκθεση και να μην αρχίσει από το μηδέν να φτιάχνει κάτι. Ξέρω ότι υπάρχει σύγκρουση στόχων μεταξύ της διαφύλαξης της επικουρικότητας αφενός και της προστασίας του καταναλωτή αφετέρου, αλλά είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε το φαινόμενο των γκρίζων ζωνών και των καταχρήσεων και καταστρατηγήσεων του δικαίου που ε, καταγράφεται σε πολλά κράτη-μέλη. Αλλά νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία και το τι είδους τόνο θα δώσουμε σε αυτή την ε, προσπάθεια, τι είδου επιλογές λέει, θα κάνουμε, γιατί καλή είναι το άνοιγμα της αγοράς, αλλά είναι μόνο μια όψη του ε, νομίσματος. Ε, θα πρέπει να κοιτάξουμε πολύ μεγάλη σοβαρότητα την καταπολέμηση των κλιματικών οργανώσεων που έχουν βρει πεδίο ελεύθερης δραστηριοποίησης, ε, εγκληματικές δραστηριότητες, ε, τις απάτες, τη διαφθορά και μόνο όταν μπορέσουμε να ε, συλλάβουμε ε, ενιολογικά όλη αυτή την εικόνα που παρουσιάζει η κατάσταση στη ψηφιακή χατοπετσικσία μπορούμε να δώσουμε τις σωστές απαντήσεις. Φερρυπίν με την αδειοδότηση, αλλά πρέπει η αδειοδότηση να είναι τέτοια ώστε να μπορεί να καταπολεμήσει τα μαύρα πρόβατα. Άρα χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα που θα εμποδίζουν τη δράση των μαύρων αυτών προβάτων, ώσπου εν τέλει να εξεφανιστούν από το πεδίο. Ευχαριστώ κύριε Σπορκέσιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή η συζήτηση που κάνουμε δεν μπορεί να αφήσει εκτός συζήτηση και γενική προϋπόθεση. Αυτή η έκρηξη των τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο ουσιαστικά είναι μια πιο μοντέρνα εικόνα των τυχερών παιχνιδιών που γινόταν στο παρελθόν σε ειδικέ όμω αίθουσε με κάποιου ελέγχου. Μπορεί να υπήρξαν και, υπήρχαν και προβλήματα στο παρελθόν, αλλά υπήρχε κάποια παρακολούθηση και υπήρχαν κάποιε ρυθμίσει, υπήρχαν ειδικοί νόμοι και υπήρχε κάποια συνειδητοποίηση κατά σας Σκεφτείτε την γαλλική νομοθεσία ενδοκιμένα για τα τεχνικά παιχνίδια. Τώρα το πανόραμα αυτό έχει αλλάξει τελώς. έχει ανατραπεί. Άλλο πράγμα και ξέραμε ότι είχαμε τις παράνομες λέσκες, είχαμε εγκληματικέ εγκληματικές πράξεις, ξέραμε ε, τι είναι παράνομο και τι, σε τι επιβάλλονται κυρώσεις. Σήμερα όμως με τη νέα πραγματικότητα των online αυτών παιχνιδιών έκανε, αν θέλετε, μια παγκόσμια μεγάλη παράνομη λέσχη όλο το διαδίκτυο. Και πιστεύω ότι και στη χώρα μου είναι πολύ ενσυχητικό το φαινόμενο και, πολύ, και παίρνει και δραματική μορφή. Αν δούμε το κύκλο εργασιών στην Ιταλία, αυτή τη δραστηριότητα μιλάμε για το 22% ε, της παγκόσμιας αγοράς στο φοντομέα. Και σκεφτείτε ότι μόνο στο 0,6% φτάνει ε, στο δημόσιο ταμείο και υπάρχει δηλαδή πραγματική φορολόγηση αυτών των δραστηριοτήτων. Σκεφτείτε επίσης την περίπτωση μιας χώρας σε κρίση, όπου 15,4 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2012 είναι ο κύκλος εργασιών. 15,4 ε, δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, από τα χέρια ποιον περνούν αυτά τα χρήματα. Έχουμε εντοπίσει 391 site που ανήκουν σε εταιρείε με 20 έδρες, κυρίως ε, Μάλτα, ε, Κύπρος, Σαν Μαρίο και ε, Γιβραλτάρ, έτσι. Έχουμε το φεστιβάλ των ε, φορολογικών παραδείσων. Και πίσω από αυτές τις εταιρείες δεν ξέρουμε ποιος κρύβεται. Μπορεί να είναι η οικογένεια Κοράλλο που ήδη πρωταγωνίστησε σε μια εξαιρετική δημοπρασία ε, για να πάρει το λότο και να πω παρενθετικά ότι στην Ιταλία το λότο ε, μας οδηγεί σε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετική. Το θέμα είναι πώς θα προστατεύσουμε τον καταναλωτή από τον εαυτό του πέρα από τις διαφημίσεις κτλ. εγώ θέλω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να το προστατεύσουμε από τους απαταιώνες αυτής της παγκόσμιας παράνομης ηλέσχης. Γιατί ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των χειρών παιχνιδιών. Να σκεφτούμε ότι αυτά τα παιχνίδια ανήκουν σε χέρια ανθρώπων που γνώμε. Δεν, γνωρίζουμε, δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό εγκληματικότητα ανήκουν αυτοί οι άνθρωποι. Ε, δηλαδή μπορεί να είναι κάποιοι κύριοι οι οποίοι χρησιμοποιούν χρήματα που μπορεί να προέρχεται και από το λαθρεπό ναρκωτικών. Ε, και έρθουν και τα ξεπλένουν αυτά τα χρήματα α, στα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο. Εκεί θα φερθούν ω κύριος, λόρδι. Όχι. Πιο πολλοί θα προσωμιάζουν όσου ε, συμμετέχουν σε εγκληματικέ οργανώσεις τύπου μαφία, ντρέκετα και ε, καμόρα. Προστασία των ανηλίκων. Πώ, τουλάχιστον οποιοδήποτε, τουλάχιστον στη χώρα μου, οποιοδήποτε μπορεί να αγοράσει μια προπληρωμένη κάρτα και να, πληρώσει, να, να παίξει συγγνώμη, ε, online χωρίς να μπορεί να διαπιστώσει κανείς αν είναι ενήλικος ή ενήλικος. Χρειάζονται πιο αυστηροί κανόνες για την εχνηλασιμότητα. Και το ποιο έχει πρόσβαση στα ε, παιχνίδια αυτά. Δεν θέλουμε διακριτική μεταχείριση σε καμία περίπτωση. Και τέλος, κλείνοντας, θα αναφερθώ σε μια άλλη ανησυχητική πτυχή που αφορά πάντοτε τη χώρα μου, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει και τι ευρωπαϊκές αρχές. Είναι κάτι που απασχολεί μόνο την Ιταλία ή όχι. Μιλάμε για παρουσία πολύ σημαντικών τραπεζικών ομίλων ε, στι εταιρείε που διαχειρίζονται αυτά τα χειρά παιχνίδια. Σκεφτείτε στη χώρα μου, έχουμε τη Μόντα και τη Σιένα που είναι στα πρωτοσέλιδα αυτή την περίοδο, αυτή η εταιρεία, η τράπεζα, συγγνώμη, για πολύ σοβαρέ εκλογικέ πράξει, μεταξύ άλλων και το ξέπλυμα χρήματο. Και συμμετέχει σε μια πολύ σημαντική εταιρεία τέτοιο του Ιχροπεθνού. Και η Intesa San Paolo, μια άλλη πολύ μεγάλη Ιταλική τράπεζα, ε, που ε, έχει το, τον έλεγχο της ΝΑΗ. Ρωτώ, είναι φυσιολογικό είναι λογικό. Οι τράπεζες. Παρότι δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στην παραδοσιακή τραπεζική δραστηριότητα της ε, ε, εξοικονόμησης χρημάτων με την κερδοσκοπία από την άλλη, ρωτώ. Αυτή η δραστηριότητα είναι λογική να απορροφούν μια οικονομική δραστηριότητα των απλών ε, ε, καταθετών που θέλουν να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα και χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα σε τόσο ύποπτες και σκοτεινές δραστηριότητες όπως είναι αυτές που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίω, εδώ πέρα δεν ε, μιλάμε για τραπεζικό κανονισμό, για τη ρύθμιση ότι αφορά τι τράπεζε ή το ξέπλυμα χρήματο. Τέλο πάντων, έχουμε 15 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μα, γιατί έχουμε και άλλο σημείο. Έχω τέσσερα άτομα στον κατάλογο μελητών. Ε, δεν ξέρω τι προτιμάτε. Ε, η Επιτροπή θα έχει και άλλη ευκαιρία να μας μιλήσει στη συνέχεια. Προς το παρόν καλύτερα να ακούσουμε τα μέλη μας. Εκτός και αν έχει κάτι συγκεκριμένο που θέλει να μας πει η Επιτροπή. Όχι, εντάξει. Τότε, καλό κύριε κύριο Φάιλερ Φίμεν, Σάρα Νουβά και Πέρες αλλά πραγματικά μέχρι δύο λεπτά το μέγιστο, γιατί θέλω να δώσω ε, το λόγο και στον εισηγητή στο τέλος, για δύο λεπτά τουλάχιστον. Θα είμαι πολύ αυστηρός λοιπόν. Αν θέλετε να κάνετε μια πιο μακροσκελή δήλωση, καλό θα το κάνετε κάποια στιγμή στο μέλλον. Βάζουμε και ρολόγια να σας βοηθήσουμε, παρακαλώ. Πολύ στόμα, Πρόεδρε. Μια και οι προτάσεις οι οποίες μέχρι τώρα έχουν διατυπωθεί με βρίσκουν απολύτως σύμφωνοι. Παραξενεύαμε που συμφωνώ και με το όσα είπε ο κύριος Κρότσμαν. Απλώς πρέπει να καταφέρουμε να κοιτάξουμε και το τι συμβαίνει στις χώρες μας. Εμείς στη Γερμανία και στα κρατήδια και στο μοσπονδιακό επίπεδο έχουμε ένα μεγάλο μείγμα νομοθεσίας ε, και πρέπει να βρούμε ρυθμίσεις ε, πιο ενιαίες. Το Σλέσφιχ Χόλστα είναι παραδείγματι, είναι μια τελείως εξαιρετική περίπτωση στην Γερμανία. Εν πάση περιπτώσει για την κυρία Μόζα και τον κύριο Κρόιτσμερ είχαμε ξαναδεί την συζήτηση αυτή. Δύο μεγάλες αλλαγές έχουν επισέλθει εντωμεταξύ. Το μεγαλύτερο δυνατό σκάνδαλο στην, στο προπό, στο ποδοσφαιρικό ε, στίχημα δηλαδή, με επιπτώσεις όχι μόνο την Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Και γι' αυτό νομίζω ότι ο κύριος Φόξ θα πρέπει να ε, ξανακοιτάξει την κατάσταση και να τη συμπληρώσει με τα πιο τελευταία στοιχεία που έχουμε δει. Ένα θέμα λοιπόν σοβαρό το οποίο επηρεάζει τον ε, φύλαθλο και πολίτη. Και το δεύτερο είναι ότι εντωμεταξύ έχει εισαχθεί η οδηγία για την για την παράνομη για την νομοποίηση παρανόμων εσόδων. Εάν συμβεί αυτό, τότε ίσω δίνουμε απάντηση και στι ε, παρατηρήσει του συναδέλφου, του Ιταλού συναδέλφου, για τι λεγόμενε ε, ε, επιχειρήσεις βιτρίνα, οι επιχειρήσεις γραμματοκιβώτιο κτλ. Δηλαδή εκεί πέρα θα εξασφαλιστεί διαφάνεια ως προς την νομοποίηση των εσόδων, χάρη στην οδηγία για την καταπολέμηση της νομοποίησης παρανόμων εσόδων. Και πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ο Φιέλνερ που είναι και ο ειδικό μας αν δεν απατώμε. Ευχαριστώ πολύ Μάλκο. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Σάλτεμόστατ ότι ε, προχωρούμε. Προχωρούμε προς τα μπρος, αλλά πολύ αργά και έχω την εντύπωση ύστερα από 9 χρόνια ότι πια δεν ηγούμαστε εμείς αυτής της πορείας, ότι απλώς προσαρμοζόμαστε σε κάποιες εξελίξεις και τεχνικού χαρακτήρα που καταγράφονται στα κράτη-μέλη. Έχει έρθει όμως πια η ώρα να πραγματοποιήσουμε ένα ακόμα βήμα και θα χρησιμοποιήσω την απαγορευμένη λέξη νομοθεσία. Νομοθεσία αλλά στο ελάχιστο εκείνο επίπεδο της προστασίας του καταναλωτή. Και προχωρώ, θα προχωρήσω και εγώ. Ε, για να πω καλά τα μονοπόλια. Καλά τα μονοπόλια. Αλλά εάν προστατεύουν τον καταναλωτή και όχι τις κυβερνήσεις και το κράτος. Και ορισμένες φορές ε, τα μονοπόλια βλέπουν να εξυπηρετούν περισσότερο τις κρατικές δομές παρά τον καταναλωτή. Σε αυτό πρέπει να δώσει απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άδειες τώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω πολλά περισσότερα θα μπορούσε να έχει πράξει για να αντιμετωπίσει την ε, γραφειοκρατική επιβάρυνση, την βραδύτητα ως προς τις άδειες, γιατί όλοι αγωνίζονται ή συναγωνίζονται καλύτερα για τον ίδιο στόχο, αλλά ε, με τρόπο διαφορετικό και άρα έχουμε τη γραφειοκρατία. Και άρα για να βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο θα πρέπει να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δράση. Η παραβάση, ο αριθμός των παραβάσεων που καταγράφονται και ο χρόνος πάνω από όλα που χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν μας ντροπιάζει. Εν τέλει, προστασία του καταναλωτή. Μου φαίνεται παράδοξο το ότι από την οδηγία για την προστασία του καταναλωτή αποκλείεται η χαρτοπεξία. Και νομίζω ότι έχουμε πολλά καλά παραδείγματα. Αλλά ή με τι άλλο, ο αυτοαποκλεισμό. Εάν αυτοαποκλείομαι από το μονοπόλιο, ναι, να αυτοαποκλείομαι και από την χαρτοπεξία. Να υπάρχει αυτή η δυνατότητα, η επιλογή. Δεν νομίζω ότι κανένα κράτο μέλο θα ερχόταν ε, ανοιχτά σε σύγκρουση με τέτοια πρόταση. Δεν θα τολμούσαν τουλάχιστον. Ευχαριστώ και πολύ χαίρομαι που σα βλέπω εδώ, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ για την ε, η παραχώρηση σας σε σχέση με το μονοπόλιο. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ και εγώ. Εν συντομία, να πω ότι είμαι σχεδόν συγγήτρια για αυτή την ε, έκθεση ε, στην Επιτροπή Πολιτισμού. Όμως εδώ βέβαια βρισκόμαστε στο πλαίσιο της Επιτροπής ΕΜΚΟ, γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο ζήτημα της προστασίας του καταναλωτή. Είναι σημαντικό να πούμε ότι τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο αποτελούν ένα σοβαρό κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ε, δημιουργία εθισμών, γιατί ε, υπάρχει πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτά από ό,τι στα παραδοσιακά τυχερά παιχνίδια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την ανακοίνωσή της Πρόκειται για μια πολύ καλή ανακοίνωση. Θα συμφωνήσω με πολλά από τα στοιχεία που παρουσίασε ο εισηγητής. Σε επίπεδο Επιτροπής Πολιτισμού ήδη είχαμε κάνει αυτή, μια τέτοια συζήτηση για αυτό το θέμα. Αναφερθήκαμε στην υπεύθυνη διαφήμιση και υπογραμμίζουμε τη σημασία των ε, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι τα παιδιά και οι ανήλικοι εν γέννη. Ίσως θα έπρεπε να υπάρξει απαγόρευση ε, των παιχνιδιών αυτών για τα παιδιά, για τους ανηλίκους και μετά για τα στημένα παιχνίδια Ήδη αναφέρθηκαν συνάδελφοι ε, σε τέτοια δίκτυα στημένων παιχνιδιών που ε, θέτει σε κίνδυνο και την αξιοπιστία του αθλήματος. Ευχαριστούμε κυρία Λιγόν Πέρες. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ένα λεπτό μόνο, γιατί ήδη υπόθεσαν πολλά. Επιμένω όμω και εγώ ότι πρέπει να επιμείνουμε πιο πολύ στην πρόληψη. Η πρόληψη είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγουμε μεγαλύτερα κακά. Ακούσαμε για μεγάλα δίκτυα για σκότεινα συμφέροντα, άρα λοιπόν χρειάζεται και διαφάνεια, πρόληψη, διαφάνεια και ρυθμίσει. Και όλα αυτά θα πρέπει να βασίσουν σε τρει βασικέ αρχέ που κατά είναι πολύ σημαντικέ. Αλληλεγγύη, τα παιχνίδια συνδέονται και με άλλες δραστηριότητε του βίου, όπως είναι και ο αθλητισμός μεταξύ άλλων, και η ακαιρεότητα είναι η γέννη. Δεύτερον, επιμείνουμε στην ανάγκη ταυτοποίηση των παρόχων των υπηρεσιών. Ο κ. Φόξ μα είπε ότι η συζήτηση και τι οργανώσει τέτοιων παρόχων υπηρεσιών και ενδιαφέρομενου φορεί και ε, μια απουσία σημείωσα ε, κάποια ένωση χριστών, παικτών, ε, ανθρώπων που έχουν φυγεί και που έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα από αυτό. Ο παίκτη πώς μπορεί να ταυτοποιηθεί ως παίκτη ή ως χρήστης. Είναι χρήστης ενός παιχνιδιού με ε, μία κάρτα και ένα τεστ ικανότητας ε, να ε, έχει αυτή τη δυνατότητα και μέχρι κάποια όρια ε, χρήση αυτών των παιχνιδιών στο διαδικτυό. Ευχαριστώ πολύ όλους σας για την τόσο πλούσια συζήτηση και σε εκπροσώπηση και πολλών χωρών σε αυτή τη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Φόξ να κάνει κάποια καταληκτικά σχόλια και να κλείσει αυτή τη συζήτηση. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Άκουσα με ενδιαφέρον όλες τις απόψεις και θα συνεργαστώ μαζί σας για να εκπονήσω μία έκθεση που ελπίζω να συμφωνήσουμε με αυτές όλοι. Και τώρα δύο λεπτά. Δεν μπορώ να πατήσω σε όλα, αλλά θέλω να σχολιάσω εντάχει το θέμα του συστήματο παιχνιδιών και του ε, ξεπλήματος των προβλημάτων. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα πρέπει να εγγυηθούμε ότι ένα καθεστώ διαδικτυακών παιχνιδιών δεν διευκολύνει αυτέ τι κλιματικές πράξει. Όμω, προσοχή, συνάδελφοι, μην ξεπερνάμε τα σκαμμένα. Ένα από τα πλεονεκτήματα, αν θέλετε, του διαδικτυακού παιχνιδιού είναι ότι αφήνει ηλεκτρονικά ίχνη. Άρα, δεν μπορεί να πει κανεί ότι στείνονται τα παιχνίδια και ξεπλένονται τα χρήματα μέσω του διαδικτύου. Ακριβώς γιατί υπάρχουν ηλεκτρονικά ίχνη που μπορούν να εντοπίσουν οι αρχές. Οπότε σας παρακαλώ να μην υπερβάλλουμε σε κάποια πράγματα. Ναι, μεν είναι όλα σημαντικά αυτά που ακούστηκαν, αλλά μην φουσκώνουμε και παραπάνω το θέμα. Και επίσης η βελτίωση προσφοράς προς το καταναλωτή. Σίγουρα πρέπει να ρυθμίσει τυχερά παιχνίδια. Συμφωνώ. Αλλά δεν πρέπει να βλέπουμε ηθικολογικά το θέμα και να το δαιμονοποιούμε. Πολλοί άνθρωποι χαίρονται, ικανοποιούνται ε, παίζοντα παιχνίδια. Ε, δεν μπορούμε στου πολιτικοί να κουνάμε το δάχτυλο και να λέμε διαφωνούμε και δεν το εγκρίνουμε. Πολύ απλά. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να φύγετε, να προλάβετε το τρένο σας, το καταλαβαίνω αλλά θα μα παρουσιάσει την έκθεση, αν κατάλαβα καλά, στις 26 Φεβρουαρίου στη Μεταγραφιστική Υπηρεσία, άρα θα εξεταστεί εδώ 20-21 Μαρτίου, 4 Απριλίου τροπολογίες, εξέταση του 20-25 τροπολογιών, ψηφίζουμε στην Επιτροπή 29 ε, 30 Μαΐου. Ευχαριστώ πολύ όλους και προσβλέπουμε σε μια ακόμη αρκετά ζωηρή συζήτηση όταν θα έχουμε μπροστά μας και την έκθεση Fox. Και πάμε τώρα στο τελευταίο σημείο για σήμερα το πρωί. Ε, με χαρά να καλωσώ στην κυρία Βερχέ. Είναι η πρώτη της έκθεση, αν δεν κάνω λάθος, στην Επιτροπή μας, ε, παρότι συμμετέχει ενεργά εδώ και καιρό εργασίες. Αξιοποιήθηκε το δίτον του υπολογιστικού νέφου στην Ευρώπη σε απάντηση ε, στην ανακοίνωση ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Ντουκατάλη είναι εδώ. Αν μπορούσαν οι συνάδελφοι να αφήσουν το χώρο ελεύθερο για να δω τον κύριο κατέλη, τον οποίο καλωσορίζουμε με μεγάλη εμπειρία, μακρά εμπειρία στα θέματα πληροφορίας. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Βερχάιν να δούμε και οι Σκιώδης, αν είναι εδώ, ο κύριος Βίγκεν Χότσα, ορθά, τα λέω, αλλά δεν τον βλέπω εδώ. Για τους ολιστές, ποιος θα μιλήσει, βρείτε τα μόνοι σας. Ο κύριος Λουκακάρτη για το Αλτή, ο κύριος Έγκστρομ, και εγώ εδώ είμαι. Αυτά. και ο επικεφαλής της Ομάδας εργασία ε, για την ε, ψηφιακή κοινωνία, αυτό αν θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ, συγγήτρια. Äh, Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, απελευθέρωση της δυναμικής του υπολογιστικού νέφου στην Ευρώπη θα έχει νόημα για να αντιμετωπίσουμε ταχύτητα της εξάπλωσης του cloud computing, αλλά και για να εξυπηρετήσουμε το σκοπό της προστασίας του καταναλωτή και να ενδυναμώσουμε τα ε, συμφέροντά του. Τι σημαίνει υπολογιστικό νέφος cloud computing, κάποιοι γνωρίζουν πολύ καλά την υπόθεση, κάποιοι λιγότερο. Λοιπόν, είναι η αποθήκευση δεδομένων βίντεο πληροφοριών σε έναν, σε έναν σερβερ σε απόσταση με τη δυνατότητα για το καταναλωτή να προσφύγει σε αυτά όταν χρειάζεται και να έχει στη διάθεσή του τα δεδομένα χωρίς να πρέπει να ε, μεταφέρει ε, μέσα στον υπολογιστή του ή σε ένα μηχάνημα τα στοιχεία αυτά. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με θέματα που άπτονται και της αποδοχής και της ε, λειτουργίας, τα κριτήρια για την λειτουργία, της ευθύνης για την απώλεια ή παραποίηση στοιχείων, την προστασία των, προσωπικών, ε, των ε, δικαιωμάτων του πνευματικού δημιουργού, όλα αυτά τα ζητήματα, νομικά ζητήματα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για να μπορεί ο χρήστης να διαθέτει στο νέφος με ασφάλεια τα στοιχεία του. και να έχει τη διαχείρισή τους, γιατί μπορεί κανείς να διαθέσει μόνος του στο δίκτυο νέφος, στο ψηφιακό νέφος τα στοιχεία του, αλλά την διαχείρισή τους ενδεχομένη και μεταφορά τους να αναλαμβάνει άλλος φορέας. Και άρα ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προστεύσει την ε, ε, διασυνοριακή πρόσβαση σε περιεχόμενα και υπηρεσίες του υπολογιστικού κράτους, ε, να προσδιορίσει τις συνθήκες για τη σύναψη των υπηρεσιών, τις συνέπειες, να εξασφαλίσει εν τέλει ένα πεδίο ασφάλειας δικαίου. Το κοινωνικό, πολιτιστικό δυναμικό που μπορεί να προσφέρει το νέφος για μένα είναι σαφές, είναι γνωστό, δεν το αφισβητώ. Μπορεί να προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για τον καταναλωτή, για τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορούν αυτές να αντλήσουν πολλά πλεονεκτήματα εφόσον μπορούν και ιδιαίτερα στις πιο απομακρυσμένες περιοχές να ε, συμβάλλουν και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Πάντως εδώ θα πρέπει να πούμε ότι προϋπόθεση για να λειτουργήσει αυτό είναι το ε, ευρυζωνικό δίκτυο, αλλιώς δεν μπορούν οι μεγάλες αυτές ποσότητες ε, δεδομένων που αναγκαστικά πρέπει να ρέουν προς το ψηφιακό νέφος να κυκλοφορήσουν κατά τρόπο ορθό ε, και αποτελεσματικό. Άρα χρειάζεται και η ευρυζωνική υποδομή. Πρέπει λοιπόν και την τεχνολογία να προαγαγούμε, αλλά πρέπει και να φροντίσουμε, να μην παρεμποδίσουμε την ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών και δυνατοτήτων χάρη στις εξαιτίας των υπερβολικών ρυθμίσεων. Εγώ επικεντρώνομαι σε ολίγα ζητήματα μόνο, το λέω ξεκάθαρα γιατί η γνωμοδότηση έχει και χρονική αλλά και ε, χωρική, χωρικούς περιορισμούς ήμουν υποχρεωμένη να περιοριστώ στα, στα περιορισμένη αυτή έκταση που έχουμε για τις νομοδοτήσεις και περιμένουμε τις τροπολογίες να κάνουμε τις σχετικές συμπληρώσεις ώστε να διατυπώσουμε ικανοποιητικά τις θέσεις της Επιτροπής μας. Επικεντρώνουμε λοιπόν αρχικά σε κάποια σημεία που είναι καταρχάς πόσο κατακαιρματισμένη είναι η ψηφιακή εσωτερική αγορά, ότι δεν είναι σαφής η όρη της χρήσης του ψηφιακού νέφους, είναι περίπλοκες οι συμβάσεις, ε, αποτρέπουν από την αξιοποίηση αυτής της υπηρεσίας των καταναλωτή, γιατί είναι περίπλοκο, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί και να επωφεληθεί των υπηρεσιών τους. Ε, Επίση, στο πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή και της επιχείρησης, για την ασφάλεια των προσωπικών του δεδομένων, των συμβάσεων, την προσέγγιση του καταναλωτή, τις κυρώσεις. Ε, και γι' αυτό θεωρώ ευπρόσδεκτη την πρόσθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συνθήκες λειτουργίας και σύναψη των συμβάσεων για το ψηφιακό νέφος με ένα σύστημα πιστοποίησης πανευρωπαϊκό το οποίο θα επιτρέπει και διαλειτουργικότητα και μεταβιβασιμότητα δεδομένων στο ψηφιακό νέφος, έτσι και η αποδοχή των επιχειρήσεων, για τις επιχειρήσεις του ψηφιακού νέφους, αλλά και για τον καταναλωτή θα διευρυνθεί, γιατί αν κανείς δεν είναι ικανοποιημένος από την υπηρεσία που του παρέχεται από ένα συγκεκριμένο πάροχο, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να πάρει τα δεδομένα του και να τα μεταφέρει σε κάποιον άλλον ε, σύνορια και η ρύθμιση των υπηρεσιών ε, του ε, νέφους επίσης είναι απαραίτητη Βήματα λοιπόν και επιλογές ε, νομοθετικού χαρακτήρα που μαζί με την αδειοδότηση θα μας επιτρέπουν ε, και την προστασία των ε, δικαιωμάτων του πνευματικού δημιουργού που ασφαλώ θα χρειαστεί, αλλά και την κάλυψη των λοιπόν εξελίξεων που μπορεί να προκύψουν με το ψηφιακό νέφος. το οποίο θα πρέπει να βρει τη θέση του ε, στην κοινωνία. Έχουμε επίσης ε, τις υπηρεσίες νέφου στον δημόσιο τομέα που μπορεί να ε, αξιοποιηθεί και να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα με λύση παραδείγματι ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η government, παροχή υπηρεσιών για τον καταναλωτή, καλύτερων ποιοτικότερων υπηρεσιών και ιδιαίτερα για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, για τους κατοίκους των πιο απομονωμένων ε, ζωνών που θα μπορούσαν ως εκ τούτου χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει φυσική παρουσία ή κτηριακή παρουσία του κράτους να εξυπηρετούνται χωρίς δυσκολία. Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο φυσικά είναι η έρευνα και η ανάπτυξη για να ενισχυθούν οι δυνατότητες, γιατί είναι τεράστιο το, δυναμικό, το αναπτυξιακό δυναμικό του νέφους και πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, καταστήσει την ανάπτυξη των ε, την ανάπτυξη σε σχέση με το ψηφιακό νέφος μία από τις προτεραιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα θα ήταν ενδεχομένω μία λύση, ώστε και να αποκτήσει περισσότερες δεξιότητες και να υποστηριχθεί ο χρήστης του νέφους, αλλά ταυτόχρονα και για να αναπτυχθούν ε, περισσότερο οι παρεχόμενες από το ψηφιακό νέφος υπηρεσίες σε συνθήκες ασφάλειας, με άρση βεβαίως των κινδύνων και ανησυχιών των καταναλωτών έτσι ώστε να βρει η Ευρώπη τη θέση της σε αυτόν τον κόσμο του ψηφιακού νέφους και να μην ε, βρίσκεται πάντοτε τελευταίος τροχός της ΑΜΑΚ σε σχέση με άλλα κράτη ή περιοχές του κόσμου που παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη και ως εκ τούτου να έχουμε τη δυνατότητα για τις επιχειρήσεις μας να δώσουμε μια όθηση για να βρουν τη θέση τους και αυτές. Μέσα στο ψηφιακό νέφος 7, όπως είπα ήταν περιορισμένη έκθεση που στη διάθεσή μου με τη γνωμοδότηση αυτή, περιμένω τις τροπολογίες των συναδέλφων, διότι ναι, έχουμε τους περιορισμούς μας και τις ε, ρυθμίσεις σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις, αλλά μπορούμε να βάλουμε και λίγο πιο πολύ ζουμί μέσα στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε δίκιο ότι σίγουρα θα υπάρχουν δυνατότητες να συμβάλλουμε και εμείς στο έργο σας. Δεν είναι κάποιος εδώ από τους σοσιαλιστές από ό,τι βλέπω για να απαντήσει. Κύριε Λεχεγκάρτ, να περάσουμε στο γύρο των ε, παρεμβάσεων των σκιωδών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την κυρία Βερχάιεν για την γνωμοδότηση. Είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανείς μαζί της για αυτό το ζήτημα. Παρότι κάποια θέματα που συνδέονται με αυτό ε, είναι ευαίσθητα σε πολιτικό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανεί με τα περισσότερα από τα συμπεράσματά τη. Ε, πράγματι, η γνωμοδότηση καλύπτει τι βασικέ πτυχέ και ιδίω ε, τι πτυχέ που αφορούν την Επιτροπή μα, δηλαδή για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Και πράγματι το απολογιστικό νέφος ε, θα μας βοηθήσει να την επιτύχουμε και να την ολοκληρώσουμε. Υπάρχουν πολλά πλέον εκτήματα από το υπολογιστικό νέφος, εξοικονόμηση πόρων, υπάρχει δυνατότητα ε, δημιουργίας θέσεων εργασίας. Βάσει μελέτης ε, του Πανεπιστημίου του Μιλάνου 1,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μάλιστα. Καθόλου αμεληταίος αριθμός σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Και βεβαίως ε, δίνει πρόσβαση σε εκατομμύρια χρήστες σε απεριόριστες πληροφορίες και δεδομένα. Και αυτό πρέπει να αντικατοπτριστεί και στη συζήτηση στον προπολογισμό, γιατί βεβαίω η σύνδεση με το διαδίκτυο είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στοιχεία. Μιλάμε για τις πλέον απομακρυσμένε περιοχές και πώς μπορούν οι κάτοικοι αυτών των απομακρυσμένων περιοχών να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έτσι, με προβληματίζει η πρόταση των κρατών μελών να κοπεί ο μηχανισμός ε, συνδέοντας την Ευρώπη. Αυτό είναι πολύ προβληματικό και ίσως θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη γνωμοδότησή μας. Όμως, προσβλέπω στη συνεργασία μου με, το, με την εισηγήτρια με τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έγκστρομ, όπως και ο προλαλής σας, θα ήθελα και εγώ να πω Οπότε και εγώ συμφωνώ με τη γνωμοδότηση. Θα ήθελα να θίξω δύο ακόμα πτυχές. Πρώτον, ε, για την επιχειρηματική κατασκοπία δεν καλύπτεται καθόλου στη γνωμοδότηση ή μάλλον στην ανακοίνωση της Επιτροπής δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Όμως, ε, η, υπηρεσία, μυστική υπηρεσία κάθε χώρα βεβαίως έχει πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα. Και τότε από τεχνική σκοπιά είναι δυνατόν κάποιος να, ε, να κωδικοποιήσει αυτά τα δεδομένα. Όμως όταν έχουμε υπολογιστικό νέφος, τότε ε, υπάρχει πρόσβαση στη μυστική υπηρεσία της χώρας. Αν δηλαδή κάποιος βάλει δεδομένα ε, σε μια χώρα, στο, ας πούμε στο Ζερμπαϊτζάν, ε, τότε η μυστική υπηρεσία έχει πρόσβαση ε, σε αυτά τα δεδομένα. Το ίδιο συμβαίνει με οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό ή όχι. Για τους περισσότερους ιδιώτες ή τις μικροβιστές επιχειρήσεις ε, δεν έχει κανένα νόημα. Αν δηλαδή οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες μπορούν να διαβάζουν όλα τα δεδομένα τους αν κάποιος έχει δηλαδή μια τοπική, μια, ε, ενέθεια τώρα της γειτονιάς. Βεβαίω, οι μεγάλε πολυεθνικέ σίγουρα δεν θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν το υπολογιστικό νεφο. Γιατί αν το κάνουν, σημαίνει ότι ε, μπορεί ακόμα και ο ανταγωνιστή σου να έχει απόλυτη πρόσβαση σε οτιδήποτε ανεβάζει εκεί πάνω. Έχει λοιπόν παρουσιάζει προβλήματα, ιδίως για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Τώρα, για τις ε, δημόσιες αρχές. Το ίδιο ισχύει. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που ε, τοποθετούνται στο ε, νέφος και μεταφέρονται σε χώρα που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά δίδεται πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν προσεκτικά. Ε, ποιες χώρες, για παράδειγμα, είναι κατάλληλες για να εξάγουμε τα δεδομένα μας. Αναφερόμαστε κάποιες φορές ε, στην ανακοίνωση για ε, τα πνευματικά δικαιώματα, όμως φαίνεται ότι κάποιοι θα θέλουν ε, τέλη για, αυτού, για αυτά τα πνευματικά δικαιώματα, όπως και για πολλά άλλα. Όμως αυτό θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για το υπολογιστικό νέφος στην Ευρώπη, για τους ιδιώτες ή τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα έμπαιναν στον πειρασμό να το χρησιμοποιήσουν. Αν υπάρχει δηλαδή φόρος μόνο και μόνο για την αξιοποίηση του νέφους, Αν δηλαδή κάποιο ε, για να βάλει κάτι στον έφο, ε, ώστε να μπορέσει ας πούμε, να ακούσει ένα τραγούδι οπουδήποτε και αν ε, ε, ταξιδέψει στην Ευρώπη, αλλά υπάρχει φόρο για την χρήση αυτή τη υπηρεσία, τότε αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Έγκστρομ. Μερικέ ακόμα προσωπικέ παρατηρήσει πριν δώσω το λόγο στου υπόλοιπου συναδέλφου. εξέτασα αυτή την πολύ καλή μελέτη που σας δείχνω εδώ. Γιατί είναι σημαντικό κάποιες τις εργασίες μας να αντικατοπτρίζονται στην πράξη. Βλέπω ότι πλέον το υπολογιστικό νέφος αφορά κυρίως τον τομέα των ε, καταναλωτών. Εγώ ήθελα να αγοράσω μια κάμερα την ε, προηγούμενη εβδομάδα. Ε, Όταν όμως συμφώνησα, τότε ο πάροχος είπε θέλετε και ένα νέφος για να αποθηκεύετε εκεί τα δεδομένα σας της φωτογραφικής μηχανής. Δεν ξέρω κατά πόσο οι καταναλωτές γνωρίζουν τους ε, όρους και οι προϋποθέσεις που συνδέονται με αυτό, αλλά πλέον γίνεται προϊόν ε, καταναλωτικό. Πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δεν λέω ότι είναι κακό σε ορισμένες συσκευέ, για παράδειγμα, όπως οι φωτογραφικές μηχανές, όπου είναι πολύ χρήσιμο να έχει κανείς έναν αποθηκευτικό χώρο ε, πέραν του υπολογιστή. Θέματα που αφορούν τις καταναλωτικές συμβάσεις και βεβαίως και την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής μας. Δεύτερον, το όλο ζήτημα της εσωτερικής αγοράς, ιδίως ό,τι αφορά πρότυπα, αλλά και τη διαλειτουργικότητα σε έναν βαθμό. Εάν δηλαδή υπάρχουν περιορισμοί ε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στον έφος ή αν υπάρχουν ε, ε, μέθοδοι κατά της ανταγωνιστικότητας κατά την παρακολούθηση κάποιων ενεργειών. Τρίτο στοιχείο που μας απασχολεί είναι ο δημόσιος ο ατομέας και οι δημόσιες προμήθειες. Ανέφερε ο κύριος Σάινστρομ ότι θα μπορούσαν κάποιες ε, δημόσιες αρχές να ε, διατηρούν τα δεδομένα μας και αν υπάρχει νομική βάση για κάτι τέτοιο. αυτό το πλαίσιο κοινής, το κοινό πλαίσιο συμβάσεων ίσως να μπορούσε να διευκολύνει την πορεία μας ε, προς ε, το υπολογιστικό νέφος. Αναφέρθηκε ότι θα υπάρχει και ένα ε, μεγάλο πακέτο για αυτό το στοιχείο και αν θα ενταχθεί στο όλο πλαίσιο πολιτικής που προωθεί η κυρία Ρέντινγκ. Σίγουρα όμως εμείς ε, προστατεύουμε όσο μπορούμε περισσότερο τα δικαιώματα των καταναλωτών. Υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, ξαφνικά εμφανιστήκατε μπροστά μου, καθυστερημένα βεβαίως. Χάσατε την αρχή, αλλά παρακαλώ έχετε το λόγο ευχαριστώ πολύ. Η στρατηγική για το ε, ψηφιακό υπολογιστικό νέφος μπορεί να έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς και γενικότερα της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς. Χαιρετίζω λοιπόν αυτές τις ε, προτάσεις. Καταγράφουν ορθήκα στην κατεύθυνση, σας έχω. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η προστασία των προσωπικών δεδομένων, την οποία θέλω να προβάλλω. Και πιστεύω ότι για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, γενικά για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, εδώ έχουμε να ε, κάνουμε με μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Και τη δυνατότητα γενικά για τις επιχειρήσεις μας να εδραιώσουν τη θέση τους σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους από την άλλη όχθη του ωκεανού. Πολλά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το ψηφιακό νέφος και που μπορούμε να αναπτύξουμε πρέπει να προβληθούν σύμφωνο με την πρόταση. Εν γέννη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και, και περιμένω να σας ξαναδούμε και σε άλλες περιπτώσεις. Ο κύριος Παπλοαριάς, κύριο Καρνόφσκι, κανείς άλλος που θέλει το λόγο. Έχουμε 10 λεπτά. Παρακαλώ να μην ε, μιλήσετε πάνω από δύο λεπτά ο καθένας. Σας, σας βάλω και το ρολόι για να σας βοηθάει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ και εγώ την Σαμπίνα, την εισηγήτρια. Εξαιρετική δουλειά ως τώρα, αν και απομένει πολύ ακόμη να γίνει. Είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία αυτή σε σχέση με το απολογιστικό νέφος. Όποιος γνωρίζει έτσι και γενικά τον όλο τομέα δεν είναι κατά. Αλλά έχω κάποια ερωτηματικά να εκφράσω. Πρέπει να μιλήσουμε για δύο ουσιώδη σημεία. Πρώτα απ' όλα, διαφάνεια και από την άλλη ασφάλεια δικαίου. Έχω αναφέρει και σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τη γνώμη μου, το υπολογιστικό νέφος είναι ένα είδος τράπεζας. Πώς είναι το τράπεζα χρημάτων. εδώ είναι μια τράπεζα δεδομένων είναι για μια τράπεζα στην ψηφιακή εποχή. Και έχω πει και σε κάποιε περιπτώσει ότι είναι και το νέο ψηφιακό νόμισμα, καθώ ε, το δολάριο είναι το νόμισμα αναφορά στις χρηματαγορές. Έτσι και εδώ, βέβαια για κάτι αντίστοιχο στην ψηφιακή εποχή τι γίνεται με την ανάκτηση των δεδομένων. Σε μια τράπεζα, όταν βάζω τα χρήματά μου, γνωρίζω πρώτα απ' όλα πού είναι. Ενώ στο, ψηφιακό, στο υπολογιστικό νέφος δεν γνωρίζω. Και όταν εγώ αποσύρω τα χρήματά μου, δεν υπάρχουν πια. Τα έχω εγώ τα χρήματά μου και έχει πλέον η τράπεζα. Με τα δεδομένα όμω, δεν ξέρω ούτε πού είναι τα δεδομένα και τα περιεχόμενά μου, κάτι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το δουλέψουμε αυτό, ούτε γνωρίζω όταν αποφασίζω να αλλάξω πάροχο, ή να τα αποσύρω και να σταματήσω να εργάζομαι με το υπολογιστικό νέφος, κρατά ή όχι αντίγραφο των δεδομένων ο πάροχος. Είναι ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσουμε. Και αν χαθούν τα δεδομένα ή τα περιεχόμενά μου, ένα πάροχο ε, που εργάζεται με τη λογική του νέφους. Χάνει τα δεδομένα μου από κάποιο πρόβλημα. Τι γίνεται με αυτά τα δεδομένα, ποιος θα με αποζημιώσει, πώς θα με αποζημιώσει κάνει μια επιχείρηση υπολογιστικού νέφους προσχωρεί σε μια άλλη επιχείρηση και ισχύουν νέοι κανόνες ή αν πτωχεύσει, αν εξαφανιστεί, αν ε, επιδεινωθούν οι υπηρεσίες που προσφέρει. Το κείμενο είναι περιορισμένο αυτή τη στιγμή, το γνωρίζω, ε, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε και όλα αυτά τα ζητήματα ώστε να αυξηθεί η αν πτωχευσει αν εξαφανιστει αν επιδεινωθουν οι υπηρεσιες που προσφερει το κειμενο ειναι περιορισμενο αυτη τη στιγμη το γνωριζω αλλα πιστευω οτι θα πρεπει να δουμε και ολα αυτα ζητηματα ωστε να αυξηθει η εμπιστοσυνη και σε αυτόν το τομέα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πρέπει να ακουστούν κάποιες καλές ιδέες και προτάσεις από αυτό. Κύριο Σασκόφσκι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι μια συζήτηση ε, η οποία θα καταλήξει να γίνει πολύ πολιτική γιατί αφορά θέματα προστασίας δεδομένων πολιτικό ζήτημα και επειδή εγώ συμμετέχω στην προσωπία με τη ΣΥΠΑ το θέμα της υποχρεωτικής ε, ε, ε μεταβίβασης δεδομένων, πρόσθεση είπα, καθαρά πολιτικό ζήτημα και αυτό και θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Όταν μιλάμε για διάφορες δραστηριότητες, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, που είναι ειδικό ο Παύλο, το θέμα του κατακριματισμου των αγορών λόγω μη ενιαία ενσωμάτωση ε, τη νομοθεσία. Άλλο πρόβλημα. Τυποποίηση και πρότυπα που είναι η δική μα δουλειά. Χωρί αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Τρίτον, αυτό που είπατε σε δημόσιες προμήθειες και ανοιχτά πρότυπα και πάλι δική μας αρμοδιότητα. Τέλος, η συζήτηση για την προστασία των δεδομένων. Αυτό που μας απασχολεί εμάς εδώ είναι η καλύτερη δυνατή προστασία δεδομένων. Αλλά πρέπει να υπάρχει ταυτόχρονα μια ισορροπία με κάποιες θεμητές ανησυχίε ε, των επιχειρήσεων να μην δολοφονούμε επιχειρηματικά μοντέλα όταν μιλάμε για την ε, ασφάλεια και τη διαφάνεια των δικτύων αυτών. Κοινοποιήσει, ε, παραβιάσει, κάνουμε Όλα αυτά θα συζητήσαμε και στα πλαίσια του νέου κανονισμού και του ψευδομένου. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ενεργοί και σε αυτό το τομέα, με ανοιχτέ και τι κεραίε. Να δούμε πώ θα επηρεάσουν όλα αυτά τα ζητήματα και το υπολογιστικό νεφος. Όλε οι μελέτε δείχνουν ότι η Ευρώπη είναι ακόμη πίσω και αν δεν δραστηριοποιηθεί δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ στου πρωτοπόρου. Υπάρχει μεγάλη ευθύνη εγώ ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για την τόσο καλή προσκευαστική δουλειά. Πρέπει όμως να προωθήσουμε αυτή τη συζήτηση, ιδίως ό,τι αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο. Αυτό το είναι πολύ γενικό. Κάποιο μπορεί να παραπλανηθεί λέγοντα ότι δεν πρέπει να μα απασχολήσει. Όχι, αντίθετα, πρέπει να μα απασχολήσει και θα πρέπει και η πτυχή τη ε, ενιαία αγορά να μπει σε αυτή τη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, τοποθέτηση και αυτή την τελευταία, αλλά και όλε. Για την δεδομένων, έχουμε ψηφίσει την ε, γνωμοδότησή μας και ε, προσέλκυσε σε μεγάλο ενδιαφέρον και θα λέγαμε πολύ καλό για την εικόνα της Επιτροπής μας. Θα δούμε ποια είναι και η θέση της ε, άλλης Επιτροπής. Τώρα πάλι το, το λόγο για λίγα λεπτά στην εισηγήτη, αλλά για λίγα λεπτά. Θα σας βάλω το ρολόι. Μήπως ξεπεράσετε τα δύο λεπτά. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε την άποψή σα. Αλλά πρώτα απ' όλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Μάλκομ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Διότι το σχέδιο κομμοδότησης αγγίζει τα μείζωνα ε, σημεία, λαμβάνοντα υπόψη ε, του περιορισμού του χώρου που δεν επιτρέπει να μπει κανεί από πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Οι συνάδελφοι εδώ έθεσαν συγκεκριμένα ερωτήματα, ανησυχίες που είχαμε και όταν εκπονούσαμε την ανακοίνωσή μας και που ενισχύσαν και τις ανησυχίες μας κατά την εφαρμογή αυτής. Και είμαστε σε αυτή τη φάση σήμερα. Αν... Ειδικά για την Επιτροπή σας, το θέμα της ευρυζωνικής ε, πρόσβασης και της πρόσβασης γενικότερα του υπολογιστικού νεύους είναι κάτι σημαντικό. Δεν αναφέρομαστε πολύ σε αυτό στην ανακοίνωση, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει καλή συμματρία και καλή ποιότητα στη, στα ευρωζωνικά δίκτυα για να μπορεί να λειτουργήσει το υπολογιστικό νέφος όχι μόνο για σταθερή πρόσβαση καθώς το πλεονέκτημα του νεύρου για τι επιχειρήσει είναι να μπορούν οι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση στις δεδομένες, τα δεδομένα συγγνώμη, όπου και να βρίσκονται. Ε, αυτό λοιπόν ήταν ένα πολύ φτωχό σχόλιο για την ενιαία αγορά και, το, και τη ρυθμιστική ατζέντα. Λέμε στην ανακοίνωση ότι υπάρχουν, έχουν δρομολογηθεί πολλέ τέτοιε ρυθμιστικέ ατζέντε και θα πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να λάβουν υπόψη και τον έφο η ψηφιακή ατζέντα, το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη δεν είναι λανθασμένο, αλλά θα πρέπει να το δούμε και υπό το πρίσμα του υπολογιστικού νεφους, γιατί αυτό είναι το μέλλον. Για παράδειγμα, αυτό που ανέφερε ο κ. Σέγκστρομ για τα τέλη που θα πρέπει να καταβάλλονται για τα αντιγραφά. Ναι. Για να μπορώ να έχω πρόσβαση τέτοια δεδομένα, α, πρέπει αυτό να συμβαίνει και με την σοφία του κυρίου Βιτορίνου την ε, διδαγματιλήσαμε από αυτά τα λεγόμενα του. Όταν, όταν έχεις άμεση πληρωμή, αυτή είναι η, η ενιαία πληρωμή και μόνο πληρωμή θα προλαμβάνεις και όχι επιπρόσθετες ε, και κατακρεματισμένες πληρωμές με τα τέλη πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει με τις επόμενε προτάσει που θα κάνουμε. Πολλά, πολλά πράγματα γίνονται ε, στην θυμιστική ατζέντα ε, και να ένα εξελίξη και θα πρέπει και αυτά να τα αμοδιοποιήσουμε και να τα εντάξουμε στη λογική του νέφους. Τώρα, πρόσβαση των πληροφοριών στις ε, ε αρχές. Πολύ σημαντικό αυτό θα ήταν υπεραπλούστευση να πούμε ότι δεν ξέρουμε πού είναι τα δεδομένα μας για το δημόσιο τομέα και για τις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν διαπραγματευτική δύναμη θα θέσουν και θα επιβάλλουν κάποιους όρους. Άρα το κρίσιμο είναι να είναι ξεκάθαρη και λεπτομερής η προσέγγιση του πώς διαχειρίζονται τα δεδομένα. Κάποια δεδομένα στρατηγικού χαρακτήρα, κάποια δεδομένα δεν έχουν καμία σημασία, κάποια άλλα έχουν μεγάλη σημασία. Χρειάζονται λοιπόν κατάλληλες λύσεις. Και να επισημάνω και κάτι που είπε η συγγήτρια. Για να επιβάλλουμε αυτές τις διατάξεις ασφαλείας θα πρέπει να έχουμε και τους δικούς μας ε, σχετικούς μηχανισμούς. Το καλό, το όφελος που δίνει τον έφο είναι η τυποποίηση όχι ότι μοιραζόμαστε το hardware, άρα η απλοποίηση πραγμάτων που στο παρελθόν απαιτούσαν ε, πολύ μεγάλη, μεγάλο κόπο για να γίνει η εξειδίκευση. Η ισορροπία λοιπόν ανάμεσα σε ένα πολύ ε, σε, μάλλον σε ένα σύστημα με επαρκές και υψηλό βαθμό προστασίας αυτό θα μπορούσε να γίνει σε επίπεδο χώρας ή παρόχου. Και εδώ τώρα προσπαθούμε να το κάνουμε από κοινού. Κάνουμε μια πρώτη προσπάθεια για να κάνουμε κάτι από κοινού, αλλά αυτή τη στιγμή κάνουμε μια καρτογράφηση προτύπων για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τεράστιο ρυθμό προτύπων που υπάρχουν. Και έτσι πιστεύω να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ε, γίνουν συνδρομητές και να πληρώνουν και αυτές τις υπηρεσίες υπολογιστή κουνέφους. Και έχω συνάδελφο εδώ από τις υπηρεσίες της ΓΔ Δικαιοσύνης, της κυρίας Ρέντινγκ. Και εδώ δουλεύουμε και αυτές τις συμβάσεις, ε, τις καταναγκαστικές που καλούνται να υπογράψουν πολλές φορές ε, οι μικροί ρεμονωμένοι χρήστες. Λοιπόν, πολλές συζητήσει που είναι εξελίξει και θέλουμε να συνεργαστούμε στενά και με την Επιτροπή σας για να καταλήξουμε ε, σε μια πολύ καλή δουλειά στο τέλος. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στην εισηγήτρια και μπορούμε να παρουσιάσουμε το χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους, για τις συστάσεις τους. Και μάλιστα τόσο νωρίς, τις ετοίμασαν. Η ε, σύνδεση με το, Euro, με το Connecting Europe Facility είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε χάρη σε αυτό το μέσο και να φέρουμε καλά αποτελέσματα. Και γι' αυτό και η κατάρτιση προγραμμάτων και σχετικών προτεραιοτήτων στον χώρο της έρευνας καταγράφτηκα τις, τις δικές μου προτάσεις προστασία των δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Έχει να κάνει άλλωστε και με τη βασική αίσθηση εμπιστοσύνη σε αυτές τις ε, υπηρεσίες. Πρέπει να γνωρίζει ο πολίτη, διαθέτω τα, ε, τα στοιχεία μου, τι τα, κάνουν, πώς τα διασφαλίζω, πώς τα προστατεύω, τι συμβαίνει σε περίπτωση απώλεια ή πόσο είναι ο κίνδυνο απώλεια. Πρέπει να προβλέψουμε λοιπόν αυτή τη διαφύλαξη με τη δυνατότητα για τη μακροπρόθεσμη και διαρκή παροχή των υπηρεσιών του υπολογιστικού νέφους, τη δυνατότητα για την μεταβίβαση, transferability και την ε, πρότασή μου θεωρώ ότι μπορούμε να την αναπτύξουμε περαιτέρω και περιμένω την πολύ καλή συνεργασία με τους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, Προθεσμία κατάθεση ε, τροπολογιών είναι 26 Μαρτίου. Έχουμε λοιπόν και το καιρό στη διάθεσή μα. Θα εξετάσουμε τι τροπολογίες στι 24 και 25 Απριλίου και θα ψηφίσουμε στι 28, 29, 30 Μαΐου. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την νομοδότησή σα. Ολοκληρώνουμε λοιπόν τα θέματα συζήτηση για σήμερα το πρωί. Σας υπενθυμίζω ότι στις 3 το απόγευμα έχουμε μια πολύ σημαντική ακρόαση εδώ, σε αυτή την αίθουσα, για την υλοποίηση της αγοράς υπηρεσιών με εξαιρετικά σημαντικούς ομιλητές. Θα σας δω λοιπόν στις 3. Πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση, επαναλαμβάνω. Καλή όρεξη.